Περνάμε στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Η προοπτική της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η διαδικασία προσχώρησης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε τώρα όλοι να καθίσουμε για να μπορέσουμε και να αρχίσουμε τις εργασίες μας. Ήδη έχουμε καθυστερήσει λίγο. Καταρχάς, θα ήθελα να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας όλους τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλωσορίσατε σε αυτή την διακοινοβουλευτική συνεδρίαση της Επιτροπής μας, της Επιτροπής δηλαδή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να καλωσορίσω εκ νέου στην αίθουσα τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια των Δυτικών Βαλκανίων και να καλωσορίσω επίσης και νέους βουλευτές, νέους ακτιβιστές, καθώς επίσης και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων που συμμετέχουν και αυτοί στη συνεδρίασή μας. Η σημερινή συνεδρίαση είναι το τελευταίο σκέλο μια υψηλόβαθμη συζήτηση στρογγυλή τραπέζη που έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων, και όπου συμμετέχουν βουλευτές από πολλές χώρες της Ευρώπης προκειμένου να συζητήσουμε μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού αναλύσαμε πριν από λίγο τη χρηματοοικονομική υποστήριξη που δίδεται προς τα Δυτικά Βαλκάνια, μπορούμε τώρα να μιλήσουμε πιο γενικά για τη διεύρυνση και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα συμφωνείτε όλοι ότι στην καθημερινή μας εργασία πολλές φορές βλέπουμε τα δέντρα και ξεχνάμε το δάσος. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγουμε κοντόφθαλμες πολιτικές κινήσεις, θα πρέπει να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας συνεχώς την γενικότερη εικόνα και τον τεράστιο μετασχηματισμό που η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση έφερε στην Ήπειρό μας. Θα πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου τις πολύ σημαντικές αλλαγές που υπήρχαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που έγινε η πρώτη σημαντική διεύρυνση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1973 μέχρι την πρώτη σημαντική διεύρυνση το 2013, όταν εντάχθηκε και η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από 15 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στο κατόφλι της μεγαλύτερης της διεύρυνσης και μετά από 15 χρόνια θα είναι εντελώς διαφορετικό το πρόσωπο πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι πεπισμένο ότι ορισμένοι συνάδελφοι από τα Δυτικά Βαλκάνια που είναι σήμερα εδώ μπορεί μια μέρα να είναι και οι ίδιοι εδώ στο Ευρωπαϊκό και φαντάζομαι ότι οι χώρες τους θα ετοιμάζονται να αναλάβουν την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ακριβώς και οι συνάδελφοι από τη Βουλγαρία θα παραλάβουν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Εστονία τον Ιανουάριο. Η ιστορία της ε, Ευρώπης ε, καταδεικνύει πραγματικά πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από τα πρώτα στάδια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην πλήρη, στην πλήρη διεύρυνση. Οι ε, βουλευτές επίσης ε, από τα εθνικά κοινοβόλια καλούνται να εγκρίνουν τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται από την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από τους νόμους αυτούς εγκρίνουν και διεθνείς ε, συμφωνίες. Ως βουλευτές, λοιπόν, όλοι δραματίζετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην έγκριση δύσκολων μεταρρυθμίσεων, προασπίζετε τα ανθρώπινα δικαιώματα, προωθείτε τις καλές ε, σχέσεις γειτονίας και συμβάλλετε στη συνέχεια της διαδικασίας της διεύρυνσης. Για μία ακόμη φορά, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σα καλωσορίσω στη μερινή μα συζήτηση. Προτού δώσω το λόγο στου ομιλητέ μα όμω, θα ήθελα να σα πω ότι έχουμε ήδη διανύμει κάρτες αγόρευση προς τους συναδέλφου βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εφόσον θέλετε να πάρετε το λόγο μπορείτε να τι συμπληρώσετε και να τι δώσετε στη γραμματεία. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο σε έναν πολύ τακτικό καλεσμένο μας εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στον κύριο Κρίστιαν Ντάνιελσον, που είναι ο Γενικός Διευθυντής για ζητήματα γειτονίας και διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της DG NEAR της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να του ζητήσω να μας κάνει μια γενική επισκόπηση της κατάστασης και ελπίζω ότι στη συνέχεια θα έχουμε μια πολύ επικοδομητική και παραγωγική συζήτηση. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση εδώ σήμερα. Κρίστιαν Ντάνιελσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευρωβουλευτές, βουλευτές ε, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα και μιλάω στην Διακοινοβουλευτική Επιτροπή. Πρόκειται για μια πολύ επίκαιρη συνάντηση και μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό της πρόοδου, αλλά να δούμε και το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον για να προχωρήσουν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή τους πορεία. Ένα βασικό στοιχείο της όλης διαδικασίας είναι η συνεργασία και η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών και βεβαίως των Πρωθυπουργών των Δυτικών Βαλκανίων. Οι χώρες έχουν προχωρήσει πολύ από το 1990 και οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, απετέλεσαν ε, κινητήριο δύναμη αυτής της μετάβασης. Βλέπουμε τα ωφέλη της απελευθέρωσης της βίζας, ε, την γενικότερη πολιτική σταθερότητα που ενισχύθηκε και επίσης... Με συγχωρείτε, τι κάνετε εκεί, λέει ο πρόεδρος. Δεν συνηθίζονται αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε την καλοσύνη τώρα να τα κατεβάσετε αυτά. Δεν ξέρω τι έγραφε εκεί, αλλά δεν συνηθίζεται εδώ πέρα και πρέπει να συμπεριφέρονται και ανάλογα οι καλεσμένοι. Έχουμε δει πρόοδο λοιπόν από τους πολέμους της δεκαετίας του 90 και η προοπτική της ε, Ένωσης ε, πετέλεσε κινητήριο δύναμη για αυτή τη μετάβαση και έχουμε περισσότερες ευκαιρίες, έχουμε περισσότερες προσωπικές επαφές, χαρακτηριστικό παράδειγμα η απελευθέρωση της βίζας και βεβαίως γενικότερα θα έλεγα όταν ε, μιλάμε για τις βελτιωμένες δημοκρατικές διαδικασίες και την πολιτική σταθερότητα και στο πλαίσιο αυτό η Σύνοδος Κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων στην Θεσσαλονίκη το 2003 ήταν ένα σημείο κάμπης για την περιοχή και οδήγησε πρώτα απ' όλα στην ένταξη της ε, Κροατίας το 2013 και τώρα υπάρχει μια νέα όθηση στην σχέση της Ένωσης με την υπόλοιπη περιοχή και τα... η σημασία των Δυτικών Βαλκανίων έχει αναγνωριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό φαίνεται και στα συγκεκριμένα παραδείγματα της ε, πρόσφατης ε, συνεργασίας μας. Ένα από αυτά είναι η μεταναστευτική κρίση, αλλά επίσης ε, και η συνεργασία μας στην παγκόσμια σκηνή. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν σαφείς και αξιόπιστες ευρωπαϊκές προοπτικές. Αυτό το έχει επαναλάβει τον Μάρτιο του 2017 φέτος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το επαναβεβαίωσε και ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης. Αλλά βεβαίως η σαφής αυτή προοπτική δεν είναι μονόδρομος. Ε, για να γίνει αυτό πραγματικότητα η βασική ευθύνη επαφίεται στις ίδιες τις χώρες. Πρέπει οι ίδιες να δώσουν πρώτη προτεραιότητα στο κράτος δικαίου, στη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι σημαντικό για τις ίδιες τις χώρες εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναφέρω λοιπόν κάποιες από τις κυρίες προκλήσεις, ξεκινώντας από το κράτος δικαίου πρόκειται για θεμέλιο όλων των αξιών ε, επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ οι χώρες έχουν κάνει σοβαρές προσπαθείς για να εξυγχρονίσουν το σύστημα της δικαιοσύνης, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα αποτελεσματικότητας και ανεξαρτησίας και λογοδοσίας. Και αυτό επηρεάζει και τα θέματα της πολιτικής στην γενική κατάσταση, αλλά είναι επίσης κάτι το οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία. Δεύτερον, ε, η μάχη κατά της διαφοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Και εδώ πέρα οι χώρες έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις του συστήματος. Υπάρχουν νέα θεσμικά όργανα. Τώρα όμως πρέπει να δούμε κάποια πολιτική δέσμευση και τα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα αποτελέσματα ερευνών, διώξεις και καταδίκες. Οι αρχές πρέπει να αρχίσουν σοβαρά να ξυλώνουν τα εγκληματικά δίκτυο, δίκτυα και να δημεύουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Το τρίτο είναι η σωστή λειτουργία των θεσμών, ειδικά των δημοκρατικών θεσμών, που είναι μια σημαντική πρόκληση. Ο κεντρικός ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων ε, πρέπει βεβαίως να έρθει στο προσκήνιο. Αυτό περιλαμβάνει και τον πολιτικό διάλογο σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα εντός του Κοινοβουλίου. Η συζήτηση πρέπει να γίνει στο Κοινοβουλίο και να προχωράει στο Κοινοβουλίο. Κατόπιν η κοινωνία των πολιτών παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και ο ενεργός ε, Διάλογο με τις κυβερνήσεις σημαίνει καλύτερες κυβερνήσεις, διαφανείς πολιτικέ διαδικασίε, λιγότερη διαφθορά και αυτοπεποίθηση στο μέλλον. Και στην διαδικασία το πέμπτο στοιχείο είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία περιέχονται στο νομικό πλαίσιο όλων αυτών των χωρών, όμως η πρακτική εφαρμογή αποτελεί ακόμα μια πρόκληση και ενώ η ελευθερία λόγου και τον ΜΜΕ παραμένει μια σημαντική ανησυχία. Τα ΜΜΕ έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν στην περιοχή ελεύθερα και ανεξάρτητα ΜΜΕ σημαίνει ότι η κυβέρνηση λογοδοτεί και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την συζήτηση και τις μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό από την πλευρά της Κομισιόν υποστηρίζουμε τις περαιτέρω πρωτοβουλίε για έναν κλάδο ΜΜΕ πλουραλιστικό και οικονομικά βιώσιμο. Το έκτο στοιχείο έχει να κάνει με την συμφιλίωση. Η μακροπρόθεσμη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην συμφιλίωση. Πρέπει να δούμε όλα τα ζητήματα που εμποδίζουν την συμφιλίωση αυτή. Έχουμε το σημαντικό διάλογο Σερβίας παιδί που αποτελεί ένα παράδειγμα. Είναι μια ιστορική ευκαιρία να βρεθεί μια μόνιμη λύση για αυτό το θέμα. Και να μην ξεχνάμε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση η ίδια ξεκίνησε μετά τον πιο καταστροφικό πόλεμο της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας, τις τάχτες της καταστροφής. Και όμως η ολοκλήρωση και η συμφιλίωση δεν σημαίνει ότι αρνούμαστε τα γεγονότα, αλλά ότι μαθαίνουμε από την ιστορία και οικοδομούμε μαζί ένα κοινό μέλλον. Αυτό ήθελαν οι πολίτες της Ευρώπης και θα έλεγα πως αυτό θέλουν και οι πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τη νέα ορμή που υπάρχει, τη νέα όθηση στις σχέσεις της Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια, για να προωθήσουμε και την συμφιλίωση αλλά και τα άλλα θέματα τα οποία ανέφερα τώρα. Στην οικονομική κατάσταση η έλλειψη ευκαιριών έχει οδηγήσει πολλούς νέους να μεταναστεύσουν ε, και επηρεάζει βεβαίως και τον ανταγωνισμό και την ποιότητα των θέσεων εργασίας και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει σιγά σιγά να περάσουμε από μια οικονομία που βασίζεται σε εμβάσματα και κατανάλωση σε μια οικονομία η οποία βασίζεται στις εξαγωγές. Και τα έχουν συμφωνήσει αυτά οι χώρες και έτσι υπάρχει ένα σωτικός χάρτης για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα που περιλαμβάνει και αναδιάρθρωση των κρατικών επιχειρήσεων και της λειτουργίας ε, του τραπεζικού τομέα. Και βεβαίως πρέπει να προχωρήσετε και στην περιφερειακή ολοκλήρωση, στη μορφή του Βερολίνου ΣΥΝ, που νομίζω ότι στηρίζει και τη διαδικασία ολοκλήρωσης για όλες τις ενλογοφόρες. Και βέβαια την ενίσχυση των χωρών μέσω έργων διασύνδεσης. Και εξυπακούεται από την πλευρά της Κομισιόν πως στηρίζουμε όλες αυτές τις διαδικασίες Έγινε σήμερα το πρωί μια συζήτηση για το προενταξιακό μέσο και θα ήθελα να τονίσω ότι πέρα από αυτό υπάρχουν επενδύσεις ε, τις οποίες στηρίζουμε για την συνδεσιμότητα, οπότε τους επόμενους μήνες θα εντείνουμε την προσπάθειά μας από την Κομισιόν και από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τώρα είναι μια σημαντική πολιτική όθηση από τις χώρες για να έχουμε αποτελέσματα στα απαραίτητα αυτά θέματα, αλλά ανέφερα και τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου και έτσι θα προχωρήσει η διαδικασία της διεύρυνσης. Το 2018 θα είναι κρίσιμο προς αυτό που τα πολλά κομισιόν επεξεργάζεται μια στρατηγική για μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία θα εγκριθεί τον Φεβρουάριο του 2018. Δεύτερον, τον Απρίλιο θα έχουμε το γνωστό πακέτο εκθέσεων που θα τεθούν επιτάπητος και θα κάνουμε μια βολιδοσκόπηση για το που βρίσκονται οι χώρες και αν μπορούν να δεχθούν Και έτσι θα έχουμε μια καλή βάση για την συζήτηση που θα γίνει τον Ιούνιο. Εν τω μεταξύ θα υπάρχει η σημαντική σύνοδος κορυφής στην Σόφια των Δυτικών Βαλκανίων την οποία αναμένουμε και βεβαίω θα είναι ένα θετικό στοιχείο στην διαδικασία. Οπότε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, είναι σαφέ ότι όλα τα θεσμικά όργανα εργάζονται προ αυτήν την κατεύθυνση και θα θέλουμε να ενθαρρύνουμε τι χώρε τη ε, περιοχή να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία αυτή και εξυπακούεται ότι θα υπάρχει συνεργασία και στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων και βεβαίως των Κοινοβουλίων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που θα παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο για να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν για τις χώρες αυτές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστούμε, Κρίστιαν Ντανιέλσον, για την αρχική σας αυτή παρέμβαση που μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση σήμερα το απόγευμα. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στους συναδέλφους από τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο καθένας από τους έξι βουλευτές έχει πέντε λεπτά το μέγιστο στη διάθεσή του. Θα δώσω λοιπόν τώρα το χρόνος στους έξι εκπροσώπους από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αλφαβητική σειρά θα ακολουθήσουμε όσον αφορά τις χώρες. Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Τάουλαντ Μπάλα. Ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά σας. Είστε Ευρωβουλευτής Επιτροπής, συγγνώμη, Βουλευτής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Κοινοβουλίου της Αλβανίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω προσωπικά για τη δέσμευσή σας για τα Βαλκάνια. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και πολλούς συναδέλφους όπως και εσάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως τον κύριο Κουκάν, τον κύριο Φλέγγενστάιν, τον κύριο Πίτουλα, τον κύριο Μποστινάρου. Συγγνώμη, δεν θα αναφέρω όλα τα ονόματα, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό το ότι παρακολουθείτε εκ του σύνεγγης τι γίνεται στα Βαλκάνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο Ταγιάννη για την στρογγυλή τράπεζα από Ξέρετε ότι ο στρατηγικός στόχος είναι βάση συνένεσης μεταξύ όλων να προσχωρήσουμε. Η πλήρης ένταξή μας στην, οικογένεια, την ευρωπαϊκή οικογένεια είναι η μόνη και η καλύτερη εναλλακτική λύση για να έχουμε δημοκρατία, ε, σωστά ανεπτυγμένη οικονομία, σωστή ε, κοινωνία και βεβαίως ασφάλεια. Έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα στο Βουλή μας για να μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή τις τάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν σχέση και με την ε, έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης. Έχουμε εγκρίνει το σχέδιο το οποίο μας ε, δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου καθορίζονται στόχοι και μέτρα για την επίτευξή τους. Η Βουλή μας, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του δικαστικού τομέα, πιστεύει ότι έχει να κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα και γι' αυτό στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων έχει ομόφωνα εγκρίνει επτά σημαντικά κλειδιά μέτρα. δέκα τρία σχέδια, πολλά σχέδια, σχέδια να μην παρουσιάστηκαν και πάρα πολλοί ε, νόμοι έχουν ε, συμπεριληφθεί και εγκριθεί σε αυτό το νέο πακέτο. Με επικοδομητικό διάλογο μεταξύ κυβέρνησης και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης προσπαθούμε να κάνουμε διάλογο και τις 17 Μαΐου του 2017 κάναμε συμφωνίες που επέτρεψαν να έχουμε πολιτική σταθερότητα. Έχει γίνει επίσης πρόοδος σε θέματα νομοθετικά, την έλεγχο της Βουλής στην κυβέρνηση, την διαφάνεια και τις διοικητικές ικανότητες και βελτίωση των ικανότητων του Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο, το οποίο έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα, διαπίστωσε ότι είμαστε ένας προορατικός και θετικός εταίρος. Συνεχίζουμε να συμμετέχουμε σε διάφορες δομές και πρωτοβουλίες στην περιοχή μας, στα πλαίσια των ε, καλών σχέσεων γειτονίας και θετικού πνεύματος. Έχουμε πάρα πολύ, ε, κάνει πάρα πολλά πράγματα για τη σταθερότητα. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις με όλες τις χώρες τις γειτονικέ στα πλαίσια πρωτοβουλειών και περιφερειακών σχεδίων. Διαδραματίζουμε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά τις δύο σημαντικές πρωτοβουλίες στα πλαίσια της συνεργασίας με τη, για θέματα νέων και για θέματα οικονομικά που θέλουν να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα, να βελτιώσουν την ανταλλαγή επαφών μεταξύ όλων και να βελτιώσουν και την ε, συμμετοχή όλων στην κοινωνία των πολιτών. Η Αλβανία συνεισφέρει με τις διάφορες ε, ε, πρωτοβουλίες της στην οικονομική σταθερότητα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι έχουν γίνει αλλαγές στην Αλβανία και από την ε, χαοτική μετακομμουνιστική χώρα που είχαμε πριν από μερικά χρόνια, σήμερα έχουμε ένα κράτος δικαίου και βεβαίως οφείλουμε πολλά για την οικονομική και τεχνική αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και τις δικές μας φιλοδοξίες να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας να γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, σεβόμενη το κράτος δικαίου και την ε, δημοκρατία. Μετά τις εκλογές μας είπαν οι πολίτες μας ότι έτσι θέλουν να είμαστε ως χώρα και είναι δέσμευση της κυβέρνησής μας να υλοποιήσει τους στόχους αυτούς. Ελπίζουμε ότι θα περάσουμε την επόμενη άνοιξη στο επόμενο βήμα ώστε να προχωρήσουμε σιγά σιγά στην πλήρη ένταξή μας στην μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Exactly Ευχαριστούμε. Τηρήσατε τα πέντε λεπτά. Έχω τώρα την τιμή να δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, στην κυρία Μποριάνα Κρίστο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα καταρχάς να σε ευχαριστήσω γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλές ε, πρωτοβουλίες έχουν λάβει χώρα και η Στρογγυλή Τράπεζα επίσης που οργανώνει δική σας επιτροπή και έχουν ως στόχο να συζητήσουμε περισσότερο την διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των ε, Δυτικών Αλβανίων. Ε, Βαλκανίων, με συγχωρείτε. Φαίνεται λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται όλο και περισσότερο με το ζήτημα αυτό. Η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα, τη σημαντικότατη θα έλεγα προτεραιότητα τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θέλουμε να διηγηθούμε σε μια κατάσταση μόνιμη ειρήνη, σταθερότητα και οικονομικού προόδου. Ήδη έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος Έχουμε υποβάλει την υποψηφιότητά μα επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λάβαμε το ερωτηματολόγιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθούμε τώρα να ολοκληρώσουμε τις απαντήσεις που θα δώσουμε στο ερωτηματολόγιο αυτό και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό πριν τα τέλη του έτους. Ένα άλλο σημαντικό βήμα είναι η έγκριση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων που οδήγησε σε διάφορα σχέδια δράσης και σε διάφορα μέτρα αλλά δυστυχώς το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είδαμε ότι δεν υπήρχε απαραίτητη πολιτική βούληση από διάφορε πολιτικέ δυνάμει, μα έχει οδηγήσει σε μια στασιμότητα όσον αφορά τι μεταρρυθμίσει και όσον αφορά την ευρωπαϊκή μα πορεία. Στην Βοσνία Ριζαγοβίνη είμαστε ενωμένοι όμω ω προ το ότι ε, θέλουμε να προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί την κοινή προοπτική όλων των πολιτικών ομάδων της χώρας. Μέχρι όμως να ευοδοθεί η προοπτική αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι από κοινού να συνεργαστούμε προκειμένου να κάνουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει επίσης να εργαστούμε προκειμένου να μεταρρυθμίσουμε την εκλογική μας νομοθεσία σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει επίσης να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την πάταξη της ε, τρομοκρατίας και της διαφθοράς. Πολύ φοβάμαι όμως ότι ε, δεν θα καταφέρουμε να σημειώσουμε γρήγορα πρόοδο όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις αυτές και θα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να διευθετήσουμε τα πιο επίγοντα προβλήματα. Επίσης, ε, δεν καταφέραμε να εγκρίνουμε μια σειρά από μέτρα που έχουν να κάνουν με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που είναι από τις απαιτήσει που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν τώρα η κατάσταση αυτή παραταθεί, δηλαδή η κατάσταση που έχει προκύψει από τον υφιστάμενο εκλογικό νόμο, αυτό σαφώ θα επιβαρύνει τη σχέση μα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σα λέω ότι ελπίζω μέχρι τα τέλη του έτου να καταφέρουμε μέσω του οικοδομητικού διαλόγου που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σημειώσουμε πρόοδο στα εκκρεμή ακόμα ζητήματα και να δώσουμε μία ικανοποιητική απάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συντοποιούμε ποια είναι τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μα, βλέπουμε και ποιε είναι οι προκλήσει που πλήττουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω για παράδειγμα η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να συνεχίσουμε τη διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ τι χώρε τη νότιο-ανατολική Ευρώπη, όχι μόνο επειδή εμεί ανήκουμε στι. Ε, χώρες αλλά επειδή και η Βοσνία Ζεγοβίνη, αλλά πιστεύω και οι υπόλοιπε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ενστερνίζονται τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουν μια μέρα να ενταχθούν σε αυτήν. Προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε σχέσεις αρμονικής γειτονίας με τις γειτονικές μας χώρες και προφανώς η διπλωματία και οι πολιτικές συμφωνίες θα πρέπει πάντα να αποτελούν την πρώτη λύση κάθε φορά που εξετάζουμε εναλλακτικέ για τη σχέση με τις γειτονικέ μας χώρες. Θεωρώ ότι έχει έρθει κατάλληλη στιγμή προκειμένου να δημιουργήσουμε μια Βοσνία Ζεγοβίνη που θα είναι τελικά ένα κράτος πλήρου ασφάλειας για όλους τους συστατικούς λαούς της χώρας μου, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθότι ένα χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης, ασφάλειας και σταθερότητας. Voilà. The next speaker is for the Assembly of Kosovo. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι των uh, Βουλών των Δυτικών Βαλκανίων, Βαλκανίων αρχίζοντας θα ήθελα να πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτή τη συνάντηση. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, διότι μας δίδει την ευκαιρία να έχουμε απευθείας ανταλλαγή απόψεων, όχι μόνο με τους αξιωματούχους των Βρυξελών, αλλά και να συγκρίνουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τις γειτονικές μας χώρες. Για μας είναι η ατζέντα, η πολιτική, πάρα πολύ σημαντική και όλες οι πολιτικές συζητήσεις έχουν σχέση με το θέμα αυτό ακόμη και όλες οι συζητήσεις που γίνονται στην Εθνική μας Συνέλευση. Δεν θα μιλήσω για τις σχέσεις μας, αλλά θα σας πω ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα. Ευθύ εξ αρχής θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει για μας μία σαφής προοπτική ευρωπαϊκής Ένωση, όπως και για τις υπόλοιπες χώρες. Όπως είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην, ε, μιλώντας για την Ένωση, ο πρόεδρος Γιούνκερ είναι στα πλαίσια της στρατηγικής της. Το Κωσυφοπαίδιο και όλες οι χώρες της περιοχής πρέπει να τύχουν αυτή τη ευκαιρία που δίδεται για να ανοίξει η προοπτική τους και να μπορέσουν να καταβάλουν προσπάθειες βελτίωσης. Το 2017 είχαμε διάφορες ε, εκλογικές διαδικασίες η τελευταία ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εκλογή. Παρά το γεγονός όμως ότι έχουμε εκλογές δεν υπάρχει αλλαγή στην δέσμευση την οποία έχουμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία ολοκλήρωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία προτεραιότητα για όλα τα θεσμικά όγαρα, κυρίως στα πλαίσια των συμφωνιών σταθεροποίησης, ανάπτυξης, αλλά κυρίως ε, και τα θέματα που αφορούν ε, την ε, Συμφωνία Σέγγεν και το θέμα των θεωρήσεων. Πρέπει να πω ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν επηρεάσει οι εκλογικές όλες αυτές τις διαδικασίες ε, την πρόοδο, αλλά παρόλα αυτά θεωρούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι θέματα προτεραιότητας. Η κυβέρνηση έχει αναθεωρήσει τις προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες μέρες ελπίζουμε ότι θα γίνει εκβαθέων συζήτηση στα θέματα αυτά και θα μιλήσουμε και θα συζητήσουμε με την Επιτροπή για τις μεταρρυθμίσεις κλειδιά που πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εμείς έχουμε αποφασίσει να, να αναλάβουμε όλες τις, ε, τα μέτρα για να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας και να συνεργαστούμε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά την απελευθέρωση για τις θεωρήσεις. Περνάει ο καιρός, αλλά είναι πάρα πολύ επίγον να ευρεθεί η λύση ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την παρούσα από το παρόν αδιέξοδο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι ε, σωστό και δίκαιο για τους κατοίκους του ε, μετά από την ε, νέα εκλογική διαδικασία υπάρχει ειδική έκθεση από ειδικού για το θέμα αυτό. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει βελτίωση και από μέρους μας υπάρχουν δεσμεύσεις ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το όλο θέμα και να εντοπιστούν τα δίκτυα τα τα οποία ενεργούν με εγκληματικό τρόπο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν οι πολίτες μας να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην θεωρούνται ως το μαύρο πρόβατο. Επίση αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις για την περιφερειακή συνεργασία με όλες τις ε, γειτονικέ μας χώρες, διότι πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι επωφελές για όλο, αν όλοι είμαστε στο ίδιο επίπεδα συνεργασίας. Ελπίζουμε ότι όλα τα προσκόμματα θα αρθούν όσον αφορά τους ε, ε περιφερειακούς ε, μηχανισμούς και τις ε, συμφωνίες. Έχουν υπογραφεί πολλά στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ των νέων και της κοινωνικότητας. Παρά κάποια προβλήματα που υπάρχουν με την μη αναγνώριση από την Σερβία και την Βοσνία Σεργοβίνη, είμαστε πεπισμένη ότι στα πλαίσια του διαλόγου που γίνεται παρά τις διάφορες εκλογικέ διαδικασίες θα προχωρήσουμε. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στον τομέα αυτό, αλλά πιστεύουμε ότι ο διάλογος θα πρέπει να γίνει με σαφές χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουν να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και όλους τα θεσμικά όργανα στι Βρυξέλλες για την υποστήριξη προς τους θεσμούς και την χώρα μας αλλά επιμένω ότι θα πρέπει να έχουμε μία σαφή προοπτική η οποία είναι σημαντική για μας και θα διατηρήσει άσβεστο τον ενθουσιασμό μας για την ευρωπαϊκή μας ένταξη. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο Σάρταν Κρούμπι, ο οποίο είναι επικεφαλή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην, στο Κοινοβούλιο τη πρώην Οικοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονία. Έχετε το λόγο. got to press the uh, Thank you. Thank you very much. Distinguished Chairman of the Committee, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε Πρόεδρε της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κύριε Ντάγγελσον, αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κοινοβουλίων των Δυτικών Βαλκανίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή, για τη διοργάνωση της συζήτησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μα συγκεντρώσατε όλους εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι εδώ πέρα, εδώ που ανήκουμε, εκπρόσωποι των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω επίση για τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω λίγο την ε, ιστορία, τη νέα ιστορία τη Μακεδονία, λέει ο την ιστορία αυτή που αποτελεί κοινή επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρχών της Μακεδονίας. Θα ξεκινήσω όμως από το 2005. Πριν από 12 χρόνια η Μακεδονία έλαβε το καθεστώς υποψήφιας χώρας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από 12 χρόνια ήμασταν κι εμείς μια χώρα που περίμενε. Το 2008 λάβαμε θετική γνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές πραγματεύσεις. Το 2009 είχαμε απελευθέρωση των θεωρήσεων θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχει υποστήριξη γι' αυτό και για το κοσυφοπαίδιο, προκειμένου να ανήκουμε όλοι τελικά στην Ευρώπη. Και τώρα, σήμερα, αν μπορείτε να φανταστείτε, έχουμε μια sui generis κατάσταση. Έχουμε μια σύσταση υπό προϋποθέσεις για την έναρξη των δεξιωτικών διαπραγματεύσεων για την πλήρη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ξεκινήσω όμως λέγοντάς σας ότι όλοι μας που εκπροσωπούμε τη δημοκρατία της ε, Μακεδονίας, ε, το κυβερνόν κόμμα και αντιπολίτευση, είμαστε δεσμε... δεσμευμένοι προς τη βασική μας προτεραιότητα, το βασικό μας στόχο, να είμαστε ανοιχτοί και διαλλακτικοί απέναντι σε όλους και η βασική μας προτεραιότητα είναι η πλήρης συμμετοχή, η πλήρης ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε μια χώρα η οποία θα αναπτύσσει καλέ γειτονικέ σχέσει με όλε τι όμορε χώρε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε συμμετέχοντα σε όλε τι περιφερειακέ πρωτοβουλίε και η Μακεδονία κατά αυτόν τον τρόπο είναι ανοιχτή απέναντι σε όλο τον κόσμο. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία εφαρμογή όλων των μεταρρυθμίσεων αυτών που έπρεπε να κάνουμε εφαρμόζοντας καταρχάς αξιόπιστες εκλογές, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές που γίνουν αποδεκτές από όλους. Και πραγματικά η φωνή των πολιτών μας ακούστηκε και αυτό ουσιαστικά αποτελούσε έγκριση για όλη τη δέσμη μεταρρυθμίσεων που έπρεπε να κάνει η Μακεδονία. Και αυτό ισχύει για όλους μας, βουλευτές, μέλη της κυβέρνησης ή τοπικού ερετού άρχοντε. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να οδηγηθούμε σε απτά αποτελέσματα για όλε τι μεταρρυθμίσει και τι ευθύνε που έχουμε αναλάβει ενώπιον σα, ενώπιον των Βρυξελών. Συνεπώς η συνέχιση της υποστήριξής σας προκειμένου να έχουμε ένα γραφείο εισαγγελέα. Έχουμε ελέξει, ελέγξει αυτή την εβδομάδα ένα νέο εισαγγελέα όσον αφορά τη Μακεδονία και έχουμε εγκρίνει μία σειρά νομοθετημάτων που έχουν να κάνουν με την προστασία των μαρτύρων, με το Δικαστικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και έχουμε προχωρήσει και σε άλλες μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το διορισμό των δικαστών, καθώς επίσης και με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την διοικητική μας νομοθεσία. Και μέχρι το τέλος του έτους θα μας σε θέση να διορίσουμε τους πρέσβεις μας και να εκλέξουμε επίσης και τους δικαστές του Σταγματικού Δικαστηρίου. Όλα αυτά τα καθήκοντα και όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι πράγματα που είχατε ζητήσει εσείς από εμά και θα έχουν όλα ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2017. Και θεωρώ ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα αποτελούν μέρος πλέον του παρελθόντος και θα έχουμε πλέον μια θετική σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μια συγκεκριμένη ημερομηνία για να ξεκινήσουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει. Προσπαθούμε παράλληλα να δημιουργήσουμε έναν επικοδομητικό πολιτικό διάλογο προκειμένου η Μακεδονία να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ζητήματα όπω η ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση, το κράτο δικαίου, η ελευθερία τη έκφραση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η καταπολέμηση διαφθορά του οργανωμένου κλίματο, οι καλέ σχέσει γειτονία και η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Όσον αφορά τι καλέ γειτονικέ σχέσει, μπορώ να σα πω ότι μέχρι τα τέλη του έτου θα είμαστε σε θέση να εγκρίνουμε στα πλαίσια του Κοινοβουλίου μας τις καλές γειτονικές μας σχέσεις με τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας πράγμα το οποίο έπρεπε να γίνει προκειμένου να επιλύσουμε και την άλλη διαφορά που έχουμε με την, τον νότιο γειτονά μας στην Ελλάδα, στο ζήτημα της, του ονόματος. Έχουμε πλέον ένα διάλογο μεταξύ της Αθήνας και των Σκοπίων και ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του 2018 θα καταφέρουμε και για αυτό το ζήτημα να βρούμε μια λύση όπως και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκα. Κάνοντας λοιπόν όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, μπορώ να σας πω ότι έχουμε ένα βασικό στόχο που πρέπει να πετύχουμε. Να ανακτήσουμε πάλι την εμπιστοσύνη όλων των πολιτών μας απέναντι στα θεσμικά όργανα της χώρας. Να καταφέρουμε να ανακτήσουμε θετικές επικοδομητικές σχέσεις με όλους τους γειτονές μας. Βλέπω συναδέλφους από τη Σερβία, την Αλβανία, το Κωσυφοπαίδιο συνάδελφοι με τους οποίους έχουμε υποδειγματικές, εξαιρετικές σχέσεις. Θα πραγματικά να τους ευχαριστήσω για την υποστήριξή τους. Εν κατακλείδη, ένα λεπτό ακόμα κύριε Πρόεδρε, να πω ε, μισό λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς εμάς. Εμείς εδώ λοιπόν στη Μακεδονία λάβαμε μια δεύτερη ευκαιρία όλοι μας πολιτικοί, πολιτικά κόμματα, κοινωνία των πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι όλες οι επιτυχίες μας είναι κοινέ ουσιαστικά επιτυχίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε πλέον μια επίσημη ημερομηνία ενταξιακών διαπραγματεύσεων Βλέπετε ότι από κοινού καταφέραμε να πετύχουμε όλα αυτά τα επιτεύγματα, συνεχίσουμε την κοινή αυτή προσπάθεια, γιατί είμαστε όλοι ενωμένοι όσον αφορά το ζήτημα της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε όλοι μια Νέα Ευρώπη. Ο κύριος Τζουγκάνοβιτς τώρα έχει το λόγο, επικεφαλής της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι πάρα πολύ καλή για την πολιτική διεύρυνση. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να εκφράσω την ευχαρίστησή μου για αυτά τα οποία είπε χτες ο κύριος Τάνοκ. Με χαρά ακούσαμε τους επένους για το Μαυροβούνιο. Θα ήθελα επίσης να τονίσω εδώ την επιστολή του κύριου Γιούνκερ όπου για πρώτη φορά έθεσε μια ημερομηνία ένταξης ε, του Μαυροβουνίου. Ελπίζουμε να είμαστε εμείς έτοιμοι. Ακόμα και πριν από την προθεσμία του 2025. Να πω επίσης ότι είμαστε υπέρ της αρχής ε, της ε, ιστιοδρομίας όπως λέγεται, ότι όποιος φτάνει πρώτος στην γραμμή θα εντάσσεται, στην γραμμή του τερματισμού και όχι στην αρχή του κομβόη. Πρέπει δηλαδή η κάθε χώρα να κρίνεται με βάση τα δικά της αποτελέσματα. Και δεν θα βοηθήσουμε κανέναν, νομίζω, εάν πληρούμε τους όρους και μετά πρέπει να περιμένουμε άλλες χώρες για να υπάρξει ένα πακέτο διεύρυνσης. Να πω επίσης ότι είμαστε υπέρ της διαδικασίας του Βερολίνου και ότι θεωρούμε ότι είναι άλλη μία μόρφη η φροντίδα που επιτυχνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Και στηρίζουμε και την διαδικασία Βερολίνο ΣΥΝ που είχε ξεκινήσει ο κ. Σίγμαρ Γκάμπριλ, ο Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, γιατί γνωρίζουμε ότι χωρίς ε, υποδομές ε, και διασυνδέσεις δεν μπορούμε να έχουμε καλές σχέσεις. Το Μαυροβούνιο δικαίως έχει αποκλειθεί πρωτοπόρος όσον αφορά την ενταξιακή πορεία. Έχουμε ανοίξει 28 κεφάλαια και τρία από αυτά έχουν προσωρινά κλείσει. Και θα ήθελα να εκφράσω την ευχαριστήσή μου για το ότι η ευρωπαϊκή μας πορεία είναι αντικείμενο συνένεσης από τους εκπροσώπους κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ε, στη χώρα μας αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Γιατί είναι τόσο επιτυχημένο το Μαυρογόνιο σε αυτή την ευρωπαϊκή πορεία. Γιατί πάντα ήμασταν μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος. Δεν είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ζούμε τις ευρωπαϊκές αξίες και θα σας πω το εξής. Γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου ήμασταν η μόνη χώρα η οποία είχε ειρήνη. Και παρά την μικρή μας έκταση δεχτήκαμε μεγάλο αριθμό προσφύγων και έτσι ακριβώς ε, επιδείξαμε το πνεύμα μας όλα αυτά σε καιρούς οικονομικής ε, κρίσης και ανακρίσεων. Πριν από 11 χρόνια ανακτήσαμε την ανεξαρτησία μας κάτι το οποίο είναι πάντα ένα δραματικό γεγονός. Και να επιθυμίσω ότι είμαστε μία από τις λίγες χώρες που έχουν πολύ καλές σχέσεις με όλους τους γείτονες, με όλους τους γείτονες μας. Επίση να πω ότι σεβόμαστε και τα δικαιώματα των μειονοτήτων εγώ. Είμαι μέλος ε, της κροατικής ε, μειονότητας του Μαυροβουνίου και οι μειονότητε, θα έλεγα ανταποδίδουν τη χάρη ε, με το να υπερασπίζονται την κυριαρχία της χώρας. Έτσι λοιπόν ζούμε τις ευρωπαϊκές αξίες και στόχος μας είναι ακριβώς να φέρουμε αυτές τις αξίες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και εδώ πέρα χρειαζόμαστε την δική σας βοήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. And last but not least, we come to Mr. Milorad Mihatovic. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Milorad Μιχάτοβιτς από το Κοινοβούλιο της Σερβίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, Με μεγάλη ευχαρίστηση λαμβάνω το λόγο σήμερα ενώπιόν σας, εξ ονόματος της Βουλής της Δημοκρατίας της Σερβίας. Πρέπει να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε παρόντες σε όλες τις συναντήσεις που προβλέπονται για την ε, συνεργασία και για την προσχώρηση της χώρας μας στα πλαίσια της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε επίσης παρόντες σε όλες τις συνεδριάσεις και όλες τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στα πλαίσια της περιφερειακής συνεργασίας, διότι καλές σχέσεις γειτονίας συνεισφέρουν στην ε, ειρήνη, στη σταθερότητα, στην περιοχή, καθώς και στην οικονομική μας ανάπτυξη. Εκτιμούμε ότι όλη η περιοχή μας θα πρέπει να αποτελέσει χώρο διαλόγου και σταθερότητας. Και αυτό είναι ένα στόχος τον οποίο νομίζω ότι όλοι θέλουμε να ελοποιηθεί και προσβλέπουμε εργαζόμενοι προς αυτό. Πρέπει να έχουμε κατά νου το γεγονός ότι από την αρχή της διαδικασίας ένταξης το 2003 σήμερα έχουμε κάποια ε, χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένες ε, ημερομηνίες. Η συνεργασία λοιπόν και οι ανταλλαγές μεταξύ όλων ημών είναι πρωτοαρχικής σημασία. Η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στρατηγικής ε, σημασίας επιλογή για την Σερβία. Και επαναλαμβάνω, πρόκειται για στρατηγική επιλογή και δεν έχουμε και άλλη επιτοχή. Θα ήθελα εντός της ε, δικής μας Βουλής να σας αναφέρω ότι υπάρχει υψηλότερο ποσοστό ε, αποδοχής αυτής της στρατηγικής μας επιλογής, σε ποσοστό 86%. Είμαστε σε διαδικασία εσωτερικών μεταρρυθμίσεων ώστε να έχουμε θεσμικά όργανα σταθερά, η οικονομία της αγοράς και θα σας πω τι έγινε μέχρι τώρα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας τέλος 2014, αρχές 2015, άρχισαν διαπραγματεύσεις για 10 κεφάλαια. Τα δύο έχουν κλείσει προς το παρόν και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος αυτού του έτους θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τρία συμπληρωματικά κεφάλαια. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, διότι από τεχνικής πλευράς και διοικητικής πλευράς η Σερβία είναι έτοιμη να αναλάβει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από όλη αυτή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Η υποστήριξη της όλης διαδικασίας ένταξης των χωρών των Δυτικών ε, Βαλκανίων εδρεώθηκε στα πλαίσια της Συμφωνίας του Βερολίνου. Για μας αυτό το οποίο είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε μέσω ε, διάφορων συμφωνιών συνεργασίας να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ε, μία από τα αρχικά μας καθήκοντα είναι βεβαίως να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής των πολιτών μας, ώστε να μπορέσουμε να αμβλύνουμε την ε, πρόβλημα εξόδου των νέων προς άλλες χώρες, όπως αντιμετωπίζετε και εσείς σε κάποιες χώρες. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να προσφέρουμε καλές συνθήκες στους νέους μας. Αυτό πρέπει να είναι μια κοινή προσπάθεια εκ μέρους όλων μας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο σημαντικά είναι τα διάφορα διακρατικά, διασυνοριακά σχέδια συνεργασίας που έχουμε στην περιοχή μας. Ξέρουμε ότι η όλη διαδικασία είναι μια διαδικασία δυτή. Αφενός η οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη, και απ' την άλλη συνεισφορά των νέων κρατών μελών με το δημοτισμό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι μπορείτε εσείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δική μας προσχώρηση να ολοκληρώσετε όλο το οικοδόμημα της ε, Ενωμένης Ευρώπης. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια να παραμείνουν ε, αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής κοινότητας στην οποία πιστεύουμε. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστούμε κύριε Μιγιάτοβιτς. Αφού ακούσαμε τις απόψεις από τους συναδέλφους των Δυτικών Βαλκανίων, περνάμε στα εθνικά μας κοινοβούλια και κυρίως στα κοινοβούλια των χωρών εκείνων που έχουν τώρα και που θα έχουν στο μέλλον την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ακούσουμε επίσης τους ευρωβουλευτές μας, καθώς επίσης και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Πάλι σας ζητώ να μην μιλήσετε για πάνω από 6-7 λεπτά. Η πρώτη ομιλήτρια, ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά σας, είναι η κυρία Κέιτ Πέντους Ροζιμάνους, η οποία είστε μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Εσθονίας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφέρατε άψογα το όνομά μου. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που διοργανώνεται σήμερα εδώ. Προέρχομαι από μια χώρα η οποία όχι μόνο έχει τώρα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και μια χώρα που θυμάται πολύ καλά όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να κάνουμε και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν πάντα εύκολος και αρμονικός. Είμαστε όμως μια χώρα που προφανώς υποστηρίζει μια πολιτική ανοιχτών θυρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μολονότι η διαδικασία μερικές φορές φαίνεται να είναι κάπως αργή, περισσότερο από ό,τι θα περιμέναμε, είναι σημαντικό να συνεχίσετε τις προσπάθειες, ακόμα και αν κάνετε μικρά βήματα, φτάνετε σιγά σιγά πιο κοντά στο τελικό σας στόχο. Τώρα, η προοπτική της διεύρυνσης θεωρώ ότι εξακολουθεί και αντιστοιχεί σε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την πρόθεση μεταρρυθμίσεων και για την πρόθεση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υποψήφιες χώρες. Και σίγουρα η ατζέντα της διεύρυνσης είναι η καλύτερη ατζέντα μεταρρυθμίσεων για τις χώρες αυτές. Οι προτεραιότητες της Προεδρίας της Εσθονίας είναι μια ανοιχτή και καινοτόμα ευρωπαϊκή οικονομία, μια ψηφιακή Ευρώπη, και μια βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Μία όμως από τις πρωταρχικές προτεραιότητές μας ήταν η ασφαλής Ευρώπη. Είναι σαφές λοιπόν ότι ε, μακροπρόθεσμα δεν μπορούμε να φανταστούμε ποτέ ότι ο ρόλος αυτός μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αρκεί να δούμε λίγο τον χάρτη της Ευρώπης για να συνειδητοποιήσουμε ότι το μέλλον των χωρών αυτών βρίσκεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων και της ευρύτερη περιοχής αποτελεί τμήμα της σταθερότητας της Ευρώπης και όπως όλοι ξέρουμε αυτό αποτελεί μέρος μιας γενικότερης παγκόσμιας σταθερότητας. Ενδεχομένως κάποιοι κάπου να είναι σε θέση να μας εξηγήσουν πώς θα μπορούσε να επιτυχήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν τα Δυτικά Βαλκάνια μέναν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ανηχώρες αυτές ξαφνικά ακολουθούσαν έναν διαφορετικό δρόμο. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ποτέ ότι τέτοιες εξελίξεις θα ήταν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν σίγουρα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ των συμφερόντων άλλων παγκοσμίων παραγόντων ενδεχομένω, αλλά όχι σαφώς υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκα επίσης σε μία διάσταση που θεωρώ ότι πρέπει να τονίσουμε λίγο περισσότερο για άλλη μια φορά η διάσταση σύμφωνα με την οποία, μάλλον η διάσταση η οποία έχει εξαφανιστεί λίγο από τις όλες τις συζητήσεις που γίνονται για τη διεύρυνση. Δεν έχει εξαφανιστεί μάλλον, αλλά δεν ε, τονίζεται αρκετά συχνά. Και η διάσταση αυτή είναι η διάσταση της ασφάλειας. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα της όλης συζήτησης και προφανώς κανείς δεν θέλει να δει την ιστορία να παραλαμβάνεται στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και σαφώ δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα σφάλματα του παρελθόντος. Έχουμε κοινέ προκλήσεις όπως η μεταναστευτική κρίση και η τρομοκρατική απειλή. Και για τους λόγους αυτούς ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε ακόμα πιο στενά, προκειμένου να καταφέρουμε να βρούμε λύσεις βιώσιμες. Η Εστονία υποστηρίζει την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περαιτέρω επέκτασή της, καθώς επίσης και το να δοθεί μια ευρωπαϊκή προοπτική στα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Και αυτό αμέριστα το έχει τονίσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα ήθελα να αφαιρθώ σε επιμέρους χώρες. Η Εστονική Προεδρία έχει προσπαθήσει να προωθήσει διαδικασία ένταξης του Μαυροβονίου και της Σερβίας και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος της Προεδρίας μας νέα διαπραγματευτικά κεφάλαια θα έχουν ανοίξει και με τις δύο αυτές υποψήφιες χώρες. Πιο συγκεκριμένα ελπίζω έως δύο επιπλέον κεφάλαια με το Μαυροβούνιο και έως τρία επιπλέον κεφάλαια με τη Σερβία. Στηρίζουμε επίσης τις εξελίξεις στην πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπου μια νέα τώρα κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στον δρόμο που οδηγεί προς μια ευρωατλαντική ολοκλήρωση. Όσον αφορά την Αλβανία, χαιρετίζουμε τη δέσμευση της υφιστάμενης κυβέρνησης να σημειώσει απτή πρόοδο σε πέντε βασικούς τομείς προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και κατά αυτόν τον τρόπο κινούνται περισσότερο προς το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων για, τα, για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη Βοσνία Ριζαγοβίνη τώρα. Ελπίζουμε ότι θα προσπαθήσει να κάνει περισσότερε μεταρρυθμίσεις, όπω και στο Κωσυφοπαίδιο, όπου η Προεδρία μα ελπίζει η νέα κυβέρνηση να κάνει περισσότερε προσπάθειες για την ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων και ελπίζουμε ότι το Κωσυφοπαίδιο θα ανταποκριθεί στι δύο προϋποθέσεις που απομένουν προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια απελευθέρωση των θεωρήσεων και ελπίζουμε να σημειωθεί περισσότερη πρόοδος στον πολιτικό διάλογο μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου που προωθείται και στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πλευράς Προεδρίας χαιρετίζουμε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική όσον αφορά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια το Φεβρουάριο του 2018. Η στρατηγική αυτή μαζί με την ετήσια δέσμη για τη διεύρυνση θα παρουσιαστεί τον Απρίλιο και κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα δημιουργηθεί μια νέα δυναμική προκειμένου να τονωθεί εκ νέου η πολιτική διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό με τη σειρά του ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσει ενταξιακέ διαπραγματεύσεις με την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και με την Αλβανία. Η Εστονική Προεδρία τονίζει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια ενεργή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίση μια στρατηγική πολιτική επικοινωνία στην περιοχή αυτή για να προβληθεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η θετική της δράση. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα άλλη μια φορά να αφαιρθώ στην εμπειρία της δικής μου της χώρας, της Εστονίας. Και να σας πω ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμούμε τις θετικές επιπτώσεις και το θετικό ρόλο που μπορεί να διδραματίσει μια φιλική θετική πολιτική ρητορική, την οποία θα μπορούσε να θετήσετε περισσότερο στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων κάθε φορά που μιλάτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι ε, η τεχνοκρατική ρητορική και μόνο δεν μπορεί ούτε να κερδίσει τους πολίτες, ούτε έχει απαραίτητα θετικά αποτελέσματα. Πέρα λοιπόν από την στρατηγική μονάδα επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωση θα πρέπει να δούμε τι λέμε και εμείς και εσείς στις χώρες σας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Χρήστο Κάτσεφ, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Βουλγαρίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Μεγάλη χαρά σας ε, μιλώ σήμερα, όχι μόνο εν ώψη της ε, Προεδρίας, αλλά και ως εκπρόσωπος ε, μιας χώρας των Βαλκανίων που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σταθερότητα και αλληλεγγύη. Οι προτεραιότητες μας λοιπόν είναι η οικονομική και κοινωνική συνοχή, η συνδεσιμότητα των ε, Βαλκανίων, η ψηφιακή οικονομία. Η Βουλγαρία αναγνωρίζει τις ευθύνε της απέναντι και στα κράτη-μέλη της ε, περιοχής αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και ο τρόπος για να υπάρξει σταθερότητα είναι να υπάρξει διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια δεν υπάρχει εναλλακτική για τα Δυτικά Βαλκάνια από το να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό οι άλλες χώρες περιοχής πρέπει να γίνουν λειτουργικές οικονομίες αγοράς που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κοινή αγοράς. Πρέπει να σεβαστούν το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνη, να καταπολεμήσουν ε, το οργανωμένο έγκλημα και να μειώσουν τη διαφθορά. Πρέπει επίσης να δείξουν ότι σέβονται τις κοινέ μας αρχές δημοκρατίας, ισότητας και ελευθερίας. Ταυτόχρονα υπογραμμίζουμε την σημασία των καλών γειτονικών σχέσεων σε ολόκληρη την περιοχή. Πρέπει το πολιτικό περιβάλλον να προσανατολιστεί προς το μέλλον των νέων γενεών. Έτσι θα δείξουμε ένα επίπεδο πολιτικής όριμότητας και βεβαίως ειδικά οι σχέσεις ε, της Βουλγαρίας ε, με την Πούγουδμού είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα για ολόκληρη την περιοχή. Βουλγαρία θα φιλοξενήσει την Σύνοδο Κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων το Μάιο του 2018 υπό την Προεδρία του κυρίου Τούσκ. Στόχος μα. θα είναι να στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα στα Δυτικά Βαλκάνια για την δέσμευση τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευρωπαϊκή του προοπτική. Και βεβαίως υπάρχει και η συγκεκριμένη εστίαση της ε, Βουλγαρικής Προεδρίας στην συνδεσιμότητα των Δυτικών Βαλκανίων. Η συνδεσιμότητα αφορά την ενέργεια, τις ε, μεταφορές, ε, την ψηφιακή συνδεσιμότητα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι λοιπόν για να ενισχυθούν οι δυσμοί εντός των Δυτικών Βαλκανίων και μεταξύ των κρατών μελών αυτή την έννοια οι χρεώσει περιαγωγή για τον κατοίκον των Δυτικών Βαλκανίων από και προ τα Δυτικά Βαλκανία ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να είναι ένα πρόβλημα. Αυτό θα αποτελέσει ένα από τα ζητήματα στην Σύνοδο Κορυφή ε, ε τη Σόφια και θα έχουμε έτσι να επιδείξουμε κάποια απτά αποτελέσματα που θα ωφελήσουν ε, τους πολίτες και των δύο πλευρών. Μετά την ομιλία του Πρόεδρου Γιούνκερ για το μέλλον της Ευρώπης απέναντι στα Δυτικά Βαλκάνια, σημειώνουμε την πρόθεση της Κομισιόν να παρουσιάσει το Φεβρουάριο του 2018 μια στρατηγική ένταξη για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Αυτό θα απαιτήσει να εστιάσουμε στα θεμελιώδη δικαιώματα, στη σταθερότητα και στην καταπολέμηση της διαφθοράς το να εστιάσουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των, θεσμών ε, της ορθής ε, διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, να μειώσουμε τους ε, κινδύνους για την σταθερότητα και είναι βεβαίως, έχει μεγάλη σημασία να βασίζεται και να κρίνεται η κάθε χώρα με βάση τα δικά της πράγματα κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής ε, Προεδρίας. Αναμένουμε τα επόμενα βήματα για τις υπόλοιπες έξι χώρες, δηλαδή νέα κεφάλαια με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Για τη Μακεδονία στηρίζουμε τις, ε, τις προσπάθειες νέας κυβέρνησης για να υπάρξουν κάποια πρώτα αποτελέσματα και να πληρώσει τα προενταξιακά κριτήρια. Είμαστε δε πεπισμένοι ότι η Αλβανία μπορεί να επιτύχει σημαντική πρόοδο τα που θα ξεκινήσουν, θα ανοίξουν τη δυνατότητα ενός πλαισίου διαπραγματεύσεων. Επίσης ε, χαιρετίζουμε το πλαίσιο διαπραγματεύσεων για την προοπτική της Βοσνίας, ε, δεδομένου και του ερωτηματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και βεβαίως ε, για το κοσφοπέδιο όπου ελπίζουμε η κυβέρνηση να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να προχωρήσουμε σε μια απελευθέρωση της ε, βίζας. Συνοψίζοντας, μιλάμε για μια στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της περιοχής και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε. Και τώρα περνάμε στον πρόεδρο της ομάδας εργασίας της Επιτροπής μας για τα Δυτικά Βαλκάνια, τον ένα και μοναδικό Έντουαρτ Κούκαν. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους βουλευτές που λαμβάνουν μέρος σε αυτή την πολύ σημαντική μας συζήτηση αυτή τη στιγμή και σε αυτό τον χώρο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να πω ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Πάντως με βεβαιότητα μπορώ να σας πω ότι η διαδικασία της διεύρυνσης όντως έχει μια νέα δυναμική θα μπορούσαμε να δούμε κάποιες θετικές αλλαγές που γίνονται σε κάποιες χώρες της περιοχής. Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εκ νέου αρχίζουν και στιάζονται περισσότερο στο ζήτημα της διεύρυνσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Και ελπίζω πραγματικά ότι οι επερχόμενες προεδρίες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην περιοχή αυτή και στις πολιτικές εξελίξεις αυτής της περιοχής. Άκουσα πολύ προσεκτικά τους προαλήσαντες από το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας, η οποία φαίνεται πλέον να είναι πάρα πολύ σοβαρή σε σχέση με την προώθηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων. Λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας τα όσα μας λέτε λοιπόν και ξέρετε ότι οι προσδοκίες και οι δικέ σα, αλλά και οι προσδοκίε των επερχόμενων προεδριών τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ ψηλέ από χώρε όπω η Αυστρία, για παράδειγμα, η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Νομίζω λοιπόν ότι οι προσδοκίε αυτέ είναι βάσιμε και ρεαλιστικέ. Σα παρακαλώ λοιπόν, προχωρήστε. Προχωρήστε στην πορεία αυτή τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πολλές εκλογές επίσης έλαβαν χώρα σε διάφορες χώρες της περιοχής. Είδαμε ότι υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν προχωρήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, δύο χώρες βρίσκονται πλέον σταθερά στη διαδικασία ένταξης και προχωρούν σταθερά με τις διαπραγματεύσεις. Έχουμε επίση θετικά μηνύματα τα οποία φτάνουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αναφέρατε πολλοί από εσά ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον λόγο του για την κατάσταση της Ένωσης, τον τελευταίο, έκανε διάφορα θετικά σχόλια για τη διεύρυνση. Τώρα, το όλο κλίμα γύρω από τη διαδικασία της διεύρυνσης είναι όλο και πιο θετικό και ελπίζω το θετικό αυτό κλίμα θα παρακινήσει και άλλες χώρες περιοχής να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις μέσα στο 2018. Παράλληλα, η διαδικασία της προσχώρησης θα πρέπει να προωθήσει περισσότερο προτεραιότητες μεταρρυθμίσεων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα παντού στην περιοχή, τα οποία θα πρέπει να ξεπεραστούν. Όλες οι χώρες δίνουν έναν αγώνα με τη διαφθορά, με το οργανωμένο έγκλημα, Πολλές φορές βλέπουμε ότι επιδεινώνεται η κατάσταση όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και κάποιες αδυναμίες όσον αφορά τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα. Προβλήματα επίσης πολιτικής φύσης όσον αφορά το κράτος δικαίου. Αυτά οδηγούν σε μία αποσταθεροποίηση, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε εκτροχιασμό της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ερχόμαστε λοιπόν στο εξή ερώτημα. Ποιες είναι οι προοπτικές της όλη διαδικασία και πώς θα πρέπει να προσεγγίσουμε την μελλοντική περίοδο που ανήκεται μπροστά μας. Ας αντλήσουμε κάποια διδάγματα από τις παρελθούσες διαδικασίες διεύρυνσης. Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα πολύ θετικό κίνητρο για το μετασχηματισμό πάρα πολλών κρατών και αυτό δεν θα πρέπει να το υποτιμούμε. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος, θα πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία ολοκλήρωσης των χωρών της, των Δυτικών Βαλκανίων και να έχουμε μεταρρυθμίσει όσον αφορά την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου θα πρέπει μόνιμα να είμαστε δεσμευμένοι απέναντι στις υποψήφιες χώρες μέσω επίσημων πολιτικών επαφών, μέσω οικονομικής υποστήριξης για, τη μεταρρυ... για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουν και μία... μέσω μιας γενικότερης εμπλοκής τους σε ευρωπαϊκά έργα, προκειμένου να υπάρχει και μια έντονη πιο έντονη ανταλλαγή μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών και πιο έντονε διαπροσωπικέ σχέσει. Είναι πολύ σημαντικό επίση να ενταχθούν οι χώρε αυτέ περισσότερο στα μεταφορικά και ενεργειακά μα δίκτυα. Να Δημιουργήσουμε επίση έναν ειδικό απεσταλμένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικό εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή αυτή. Βέβαια, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μια διαδικασία αμφίδρομη, όπω ακούσαμε όπως εμείς δεσμευόμαστε απέναντι στις χώρες των Δικών Βαλκανίων, έτσι και αυτές θα πρέπει να δεσμεύονται για τις μεταρρυθμίσεις και τις βασικές αξίες. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες, αντιμετωπίσαμε πολλές κρίσεις που εμποδίσουν τις προοπτικές διεύρυνσης ορισμένων χωρών που έχουν οδηγήσει επίσης σε εσωτερικές πολιτικές κρίσεις που έχουν να κάνουν με αδυναμίες όσον αφορά τους δημοκρατικούς θεσμούς όσον αφορά το κράτος δικαίου ή πολλές φορές με καθεστώτα τα οποία ε, έχουν μια πολιταρχική διάσταση. Ξέρετε ότι ε, αυτά οδηγούν πολύ συχνά σε γενικότερη αποσταθεροποίηση, ε, μποϊκοτάρουν πολλές φορές τη διαδικασία της διεύρυνσης και μπορούν να την εκτροχιάσουν και εντελώ. Δεν θα αναφερθώ τώρα συγκεκριμένα σε χώρες, ξέρετε σε ποιες αναφέρομαι. Ξέρετε ποιες εννοώ. Προκειμένου λοιπόν να σημειώσουμε πρόοδο, θα πρέπει να ανανεώσουμε τις δεσμεύσεις μας και εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα πρέπει ξεκάθαρα να θέσουμε σαφείς στόχους και θα πρέπει για άλλη μια φορά η διεύρυνση να αποτελέσει σημαντικότατη προτεραιότητα του πολιτικού θεματολογίου μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. ευχαριστούμε, κύριε Έντουαρτ Κούκαν. Και θα ήθελα να τονίσω πόσο εξαιρετική δουλειά έχετε επιτελέσει μέσω του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Και τώρα θα δώσω το λόγο της, στην αναπληρωτή διευθύντρια ε, υπεύθυνη για θέματα Ευρώπης και Αντρικής Ασίας, την Αντζελίνα Άισχορτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που είμαστε όλοι εδώ. Βλέπουμε να υπάρχει σύγκληση απόψεων σε πολλά θέματα. Θα ήθελα να αναφερθώ, αν μου επιτρέπετε, σε τρία θέματα. πρώτα απ' όλα, Θα ήθελα να αναφερθώ στα νέα κεφάλαια που μας απασχολούν. Την ασφάλεια, το μεταναστευτικό, την ε, σφαιρική στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκανία που εισήγαγε η κυρία Μογκερίνη και ένα νέο κεφάλαιο, μια νέα φάση στο διάλογο, μια νέα δυνατότητα που ε, δόθηκε στα πλαίσια της νέας στρατηγικής έτσι, για του χρόνου, έτσι όπως ανέφερε ο, ο πρόεδρος ε, Γιούνκερ όταν μίλησε το μέλλον της Ένωσης. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές νέες δυνατότητες και ακούσαμε ότι ευθυγραμμίζονται προς και η παρούσα και η επόμενη Προεδρία. Βεβαίω όλα αυτά να συνοδεύονται με σοβαρή εργασία. Επίσης πρέπει να πω ότι τα κράτη-μέλη και τα κοινοβούλια και όλοι εσείς ενεργείτε βάσει της βούλησης των πολιτών σας. Εάν δούμε ποια είναι η υποστήριξη για περαιτέρω διεύρυνση, Έχουμε ποσοστά 35 με 45% πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και βλέπουμε ότι στις ίδιες τις χώρες των Βασκανίων έχουμε μεγάλο ποσοστό υποστήριξη στην Αλβανία, 86%, το υψηλότερο στη Σερβία 49% το χαμηλότερο, αλλά εδώ βλέπουμε ότι είναι μισογεμάτο το ποτήρι και έχουμε ακόμη χώρο βελτίωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει η κοινή γνώμη να βελτιώσει την ε, πεσοστά αυτά. Και χαίρομαι που σήμερα μπορούμε να κάνουμε κάτι, διότι έχουμε πάρα πολλούς νέους μεταξύ μας. 25% συμπεριλαμβανομένου και του κύριου Φλάκενστάιν, 25% των ε, λαών των Βαλκανικών χωρών γεννήθηκε μετά από το 90, 1990 και κάποιοι από εμά επίσης ή από εσά. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να προσβλέπουμε προς το μέλλον. Στις νέες γενιές με τις οποίες θα πρέπει να εργαστούμε και να αποδείξουμε και εμείς οι αξιωματούχοι, τα μέλη των κοινοβουλίων και όλοι ότι μπορούν οι βουλές παντού να λειτουργήσουν σωστά και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίας. Υπάρχουν βεβαίως κάποια θέματα εκκρεμή ακόμα όσον αφορά τα θέματα λειτουργίας των Εθνικών Βουλών. Πρέπει όλοι αυτό να το έχουμε ε, κατά νου. Ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος της κάθε Βουλής σε σχέση με τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά ξέρουμε ότι θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες ακόμη για να είμαστε σίγουροι ότι όλοι γνωρίζουν προς τα που θέλει να στραφεί η χώρα της προς το μέλλον. Ελπίζω ότι στους επόμενους έξι μήνες με στα πλαίσια της συνεργασίας θα παρουσιάσω ε, σε όλους εδώ εκ μέρους υπηρεσίας μας με την κυρία Μαγκερίνη ε, πολλά θέματα στα οποία θα έχει επιτευχθεί πρώτος για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα η προσχώρηση. Ευχαριστούμε, Αντζελίνα Άιχορστ. Ακούσατε όλους τους ομιλητές εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων και της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου. Τώρα έχουμε χρόνο για απαντήσεις και ερωτήσεις. Προς το παρόν. Έχουν ζητήσει το λόγο 16 συνάδελφοι. Θα ήθελα να προτείνω κατανότα το όριο 3 λεπτά χρόνο ομιλίες για τον καθένα. Αρχίζουμε με τον Κνούκ Βελσνστάιν, ο οποίο είναι εισηγητή για θέματα που την... Ευχαριστώ, θα μιλήσω γερμανικά. Δεν ξέρω πώς τα πάτε εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά εγώ έχω εντύπωση ότι όλα αυτά τα έχω ξανακούσει που ακούσαμε σήμερα. Γι' αυτό θα είμαι σύντομος. γνωρίζουμε όλοι ότι αρκεί μια ματιά στο χάρτη για να διαπιστώσουμε ότι οι χώρες ε, των Δυτικών Βαλκανίων είναι στο κέντρο της Ευρώπης ούτως ή άλλως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να δείξουμε ως ευρωπαϊκά θεσμικά Οργάνωση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θέλουμε αυτές τις χώρες γιατί ο χρόνος που χρειαζόμαστε για να διαπραγματευτούμε, για να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις είναι μεγαλύτερος ε, από όσο νομίζαμε. Και εμείς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μην μετατρέψουμε την ε, διαδικασία αυτή σε ένα γραφειοκρατικό, τεχνοκρατικό τέρας και να περιοριστούμε στα απλά πράγματα. Δεν νομίζω κανένα στο Βελιγράδι, για παράδειγμα, να ξέρει τι σημαίνει ένα κεφάλαιο. Δεν χρειάζεται λοιπόν τόσο κήρυγμα και καλό είναι να κοιτάξουμε και τη δικιά μας την πλευρά. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν ε, γρήγορα και τα χαρτιά μένουν και πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη. Ναι, ωραία, συμφωνώ. Αλλά τι πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, να επιδείξει μεγαλύτερη συνέπεια. Οι νέοι που τους είπατε δεν επιτρέπεται το χαρτί, κρατούσαν ένα χαρτί που έγραφε απελευθέρωση βίζας για το κοσμοπέδιο. Αυτό έγραφε. Και συμφωνώ και εγώ μαζί τους. Πρέπει να πιέσουμε να συμβεί αυτό, γιατί μια χώρα η οποία εντάξει έχει το χύψη πρόβλημα, ε, βρίσκεται στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ πέρα έχουμε κάποιες ε, χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζουν πλήρως τα του κανονισμού των συνόρων. Η ΔΕ Αλβανία έχει κάνει πολύ περισσότερα στις μεταρρυθμίσεις των τομέα της δικαιοσύνης από κάποια μέλη. Γι' αυτό είναι λάθος ο πρόεδρος της Κομισιόν ε, να αναφέρει μόνο κάποιες χώρες ε, ότι θέλουν μεταρρυθμίσεις και όχι κάποιες άλλες. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Προτελευταίο. Πρέπει να δείξουμε ότι θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και η ε, απελευθέρωση της βίζας θα είναι κάτι το απτό, κάτι το οποίο θα έχει ο κόσμος. Στο ακριβώς θα πρέπει να δούμε το θέμα αυτό του roaming ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μα, από αυτό κερδίζει και ο επιχειρηματία ε, και οι νέοι και πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά. Τελευταίο. πρέπει να πούμε και στους ε, ψηφοφόρους μας ότι είναι σημαντικό να έρθουν σε εμάς οι άνθρωποι και τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, όχι απλά να ζουν δίπλα μας. Αν δεν τους το πούμε, δεν θα πιστούν και οι δικοί μας οι ψηφοφόροι. Αν λοιπόν θεωρούμε πράγματι ότι είναι μια σχέση η οποία είναι αμοιβαίως υποφελή, ε, πρέπει να το λέμε και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σε ευχαριστώ. Vielen Dank, lieber Kollege Knut Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. Περνάμε τώρα στου προσκεκλημένους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και νομίζω ότι σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να είναι η Ιταλία γιατί βεβαίως ε, συμβάσχουμε με τον πόνο σας, ε, με τον πόνο του αποκλεισμού από το παγκόσμιο κύπελο. Η κυρία Μαριέτα Τιντέη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν τα ξεκινάμε καλά τα πράγματα, λοιπόν, θα πάμε λίγο καλύτερα στη συνέχεια. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, αλλά και τον ε, Επίτροπο Χάν που είναι υπεύθυνο για τα ζητήματα διεύρυνσης και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την γραπτή απάντηση που έδεσε σε σχέση με μια ερώτηση που υπέβαλε η δική μας η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Θέλαμε ουσιαστικά να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία της διεύρυνσης θα παραμείνει αξιόπιστη, γιατί η αξιοπιστία αυτή ουσιαστικά διαμορφώνει τις σχέσεις μας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς επίσης ε, αποτελεί προϋπόθεση για τον εξεχρονισμό των χωρών αυτών αν μία χώρα ξεκινά μεταρρυθμίσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει συνεχώς την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να δούμε καταρχάς ποια θα είναι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η δέσμευση των ίδιων των ε, κρατών της περιοχής εκείνης, όπως είχαμε δει στην περίπτωση της Κροατίας. Είναι σημαντικό να μην λαμβάνουν οι χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια αρνητικά, αποθαρρυντικά μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερη αποσταθεροποίηση της χώρας και της ευρύτερη περιοχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης τα όσα υπόθηκαν στην επιστολή αυτή για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να λάβουν χώρο όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, την οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με τα κριτήρια της Κοπεχάγης και της Μαδρίτης. Ας μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να επηρεάσουμε περισσότερο την κοινωνία των πολιτών στις χώρες αυτές προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τα θετικά ωφέλη της διεύρυνσης και της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι η δέσμευση της Ιταλίας όσον αφορά τη διάσκεψη που έλαβε χώρα στην Τεργέστη τον Ιούλιο που μιλήσαμε για ζητήματα όπως οι επενδύσεις, η ενέργεια, οι μεταφορές. Στην Τεργέστη ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τις μεταφορές προκειμένου να δημιουργηθεί μια περιφερειακή ολοκλήρωση επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών. Όπως είπε και ο Επίτροπος Χαν, αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εναλλακτική της διεύρυνσης, αλλά προωθεί περισσότερο την προοπτική της διεύρυνσης. Σε σχέση λοιπόν με αυτό το ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί συνεχώς από πολιτικής πλευράς, είναι πολύ σημαντικό η μελλοντική βουλγαρική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τονίσει τα συμπεράσματα της διακοινοβουλευτικής διάσκεψής μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι στα πλαίσια της διάσκεψης αυτής έχουμε ίσως τα μόνα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή για να ελέγχουμε περισσότερο την πρόοδο στις χώρες αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε στα πλαίσια των πορισμάτων των διακοινοβουλευτικών αυτών συνεδριάσεων πώς αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως η διεύρυνση και οι μεταρρυθμίσεις των Δυτικών Βαλκανίων. Από το 2016 και μετά, μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία και σε σχέση με την στάση έπειτα του Ερντογάν και τη γενικότερη στάση της Άγκυρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι η επιρροή της Τουρκίας και επιπτώσεις από, την εξέλιξη, από τις εξελίξεις αυτές στα Δυτικά Βαλκάνια. Ας μην ξεχνάμε ότι η ευημερία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων εξαρτάται από την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό οι χώρες αυτές να αισθάνονται ασφαλείς και να μπορούν να αντιμετωπίσουν εξωτερικές, απειλέ απειλές η τρομοκρατία ή ανεξέλεγκτη προσφυγική κρίση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζητήματα όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η σταθερότητα επηρεάζονται από όλε αυτές τις εξελίξεις. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι οι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν πάρα πολύ από πολιτικής και οικονομικής πλευρά στι χώρες αυτές και πολλές φορές εις βάρος του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε τώρα τον πρώην Υπουργό Συνάδελφο από την Κροατία, Μύρο Κόβατς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ντέιβιτ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα στις Βρυξέλλες και μπορώ να μιλάω σε εσά για τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας. Πρώτα απ' όλα είναι ενθαρρυντικό το ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ ανέφερε στην ομιλία του Ιντομένου της Ένωσης τα Βαλκάνια και είπε «Εάν θέλετε περισσότερη σταθερότητα στην γειτονιά, μου, θα πρέπει να έχετε μια προοπτική αξιό... πρέπει να έχουμε μια προοπτική αξιόπιστη προς τους γείτονες των χωρών αυτών. Πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό. Και φέτος πρέπει να πω ότι σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων έχει συζήτηση για τα Δυτικά Βαλκάνια μετά από 7 χρόνια, δεν με απατά η μνήμη μου. Συμφωνώ λοιπόν πλήρω με τον κύριο Φαλκενστάιν και με την δική σου συλλογιστική, Ντέιβιντ ότι τα Δυτικά Βαλκάνια είναι στο μάχη της Υπήρου μας. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να το φροντίσουμε το κομμάτι αυτό της Ευρώπης. Θα πρέπει να είμαστε η κύρια κινητήρια δύναμη και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε άλλες εξωτερικές δυνάμεις να είναι πιο δυναμικές από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε περισσότερο τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Εάν δείτε την όλη περιοχή, θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι. Έχουμε το θέμα μεταξύ Βοσνίας Σκοβίνης και Σερβίας, το θέμα μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα, πρόβλημα μεταξύ της Αλβανίας και της Μακεδονίας, λέει ο μιλητής. Υπάρχουν ε, πιθανότητες τρομοκρατικών επιθέσεων και όπως προαναφέρθηκε υπάρχουν πρώην μεγάλες δυνάμεις οι οποίες κάνουν στην περιοχή αυτή κάποιους υβριδικού τύπου πολέμους. Η Κροατία είναι η πρώτη χώρα η οποία επιτυχώς ολοκλήρωσε όλη τη διαδικασία. Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος, είναι δυνατόν να αλλάξει μια χώρα για να αποτελέσει μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλει μία σημαντική προσπάθεια συμφιλίωσης, όπως και άλλοι εκτός Ευρώπης το επιθυμούν. Θα πρέπει στα πλαίσια λοιπόν ενός επικοδομητικού διαλόγου να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ίσως δημιουργούν τα προβλήματα και έτσι να βρεθεί λύση γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε την όλη διαδικασία ένταξης. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής από τη Γαλλία, η κυρία Λιλιάνα Τόγκη. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να δηλώσω εδώ πόσο προσελωμένη είναι στο στόχο αυτό της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων η Γαλλία. Το είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Μακρό στην Σορβόνη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε, να ανοίξει προς τις χώρες των Βαλκανίων όταν θα είναι έτοιμες να σεβαστούν πλήρως το κεκτημένο, το κοινωτικό κεκτημένο και την δημοκρατία. Θα ήθελα να πω ότι οποιαδήποτε βήματα προς την ε, ένταξη θα πρέπει να γίνουν όταν όλα τα κριτήρια πληρούνται. Θέλουμε να γίνει μία σωστή περαιτέρω διεύρυνση, αλλά με σοβαρότητα και σεβασμόλης της ε, διαδικασίες. Παρά το γεγονός ότι πρόσφατα έχουμε πολλές θετικές εξελίξεις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, υπάρχουν σημαντικά κενά και προβλήματα, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι προηγουμένω. Είμαστε όμως αισιόδοξοι. Ξέρουμε ότι οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών θέλουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις και θα θέλαμε τα λόγια να συνοδευτούν από έργα συγκεκριμένα και από μεταρρυθμίσεις οι οποίες πραγματικά θα τεθούν σε ισχύ. Χαιρετίζω τις πολύ ενθαρρυντικές ε, προόδους που έχουν γίνει στην ε, διαδικασία ένταξης Μαυροβουνίου και Σερβίας, θα ήθελα ολοκληρώνοντας επίσης να έχω κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά το χρονοπρόγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής ώστε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και την πρώην Δημοκρατική ε, engagée aux côtés des pays. Δημοκρατία ε, Ευχαριστώ. Merci, madame. Ευχαριστώ πολύ. From the European Parliament, Mr. Epitideos. Να μου τώρα στον κύριο Επιτίδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στις προσπάθειες που καταβάλουν οι χώρες τους να ξεπεράσουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και να γίνουν ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα ήθελα να απευθύνω δύο ερωτήσεις στον εκπρόσωπο της Αλβανίας. Ε, είπατε προηγουμένως ότι ένα από τα στοιχεία τα οποία έχει βελτιώσει η χώρα σας έχει σημειώσει επιτυχία είναι οι σχέσει καλή γειτονία με τι ε, γειτονικέ χώρε. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αυτό επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι δεν ισχύει. Η χώρα σας εγείρει εδαφικέ αξιώσει κατά τη ε, περιοχή τη Υπήρου, η οποία καλείται τσαμουριά και επίση, εδώ και πολλά χρόνια παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα τη ελληνική μειονότητα τη Βορείου Υπήρου που κατοικεί στο νότιο τμήμα τη χώρα σα. Παρεμβαίνει στις ε, εκλογές κατά τρόπο ο οποίος δεν είναι αποδεκτός και επίσης δεν αποδέχεται να αποδώσει τις περιουσίες τους στους ανθρώπους της μειονότητας. Πρόσφατο παράδειγμα είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται με νομότυπα τεχνάσματα να αφαιρεθεί η περιουσία από τους κατοίκους της Χιμάρας. Τέλος, παραβιάζει και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα των θρησκευτικών ελευθεριών. Γκρέμισε το καλοκαίρι την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου στις Ρημάδες, συγγνώμη του Αγίου Θανασίου στις Ρημάδες και τώρα επιβάλλει εισιτήριο στους πιστούς για να μπουν στις εκκλησίες. Θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι δείγματα καλής γειτονίας. Και η δεύτερη ερώτηση, για ποιο λόγο η χώρα σας θέλει να κάνει συνομοσπονδία με το κοσυφοπέδιο. Ευχαριστώ. Thank you. We come to... Σας ευχαριστώ. Ερχόμαστε στον κύριο Ρισάρ από την Πολωνία. Ας είστε. μιλήστε απευθείας θα έλεγα με τον Έλληνα συνάδελφο. Καλό είναι νομίζω να μιλάει κάποιος από τη Χρυσή απευθείας με τους Αλβανούς. Ερχόμαστε στον κύριο Ρίσαρ Μάιερ. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. μπορούμε να συζητήσουμε για τα Δυτικά Βαλκάνια με τους υπόλοιπους εδώ συναδέλφους. Κυρίες και κύριοι, η Πολωνία είναι σαφώς υπέρ της πολιτικής ανοιχτών θυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της διεύρυνσης μπορούμε να οδηγηθούμε σε μεγαλύτερη ασφάλεια, σταθερότητα, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και θετικές αρμονικές σχέσεις γειτονίας στα Δυτικά Βαλκάνια και η ίδια η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται από την ασφάλεια αυτής της περιοχής. Η περιοχή αυτή είναι μέρος της Ευρώπης και συνεπώς οι φίλοι μας από τις χώρες Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να ενταχθούν συντομότατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας δούμε το ζήτημα των Δυτικών Βαλκανίων από μια διαφορετική οπτική γωνία. Μετά τη μεταναστευτική κρίση, μετά την κρίση του Brexit, οι πολίτες πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιμένουν να δούνε μια κάποια επιτέλους επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αποδεχθούμε τους κατοίκους των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως πραγματικά να πετύχουμε αυτή την θετική εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι η προσχώρηση των κρατών αυτών θα οδηγήσει στον εξυγχρονισμό των κρατών αυτών, στον εκδημοκρατισμό τους στην τήρηση των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών, αλλά θα καταφέρουμε και εμείς, οι ήδη φυστάμενοι αν θέλετε πίκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξυγχρονιστούμε εκ των έσω χάρη στην παρουσία των νέων αυτών πολιτών. Ενθαρρύνω λοιπόν του συναδέλφου από τα Εθνικά Κοινοβούλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενθαρρύνουν του συναδέλφου μα από τα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Μπορούμε ερχόμενοι σε επαφή με του ανθρώπου αυτού, με του συναδέλφου, να μοιραστούμε τη σωρευμένη εμπειρία που έχουμε από την ένταξη και τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα η όλη αυτή διαδικασία δεν είναι απλώ μια γραφειοκρατική, τεχνοκρατική διαδικασία ο κύριος Κρίστιαν Τίμπριν Γέντε, το αρχιτολόγο από την Νορβηγία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι εξελίξεις στην περιοχή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικές για όλους μας. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί και η κοινωνική και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας αυτής οι, κοινωνι... τα... κοινωνικές προκλήσεις, η οικονομική ανάπτυξη και όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να επιληθούν και η προοπτική της συνεργασίας στα πλαίσια της Ευρώπης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Για πάρα πολύ μεγάλο, εδώ και πάρα πολύ καιρό εμεί υποστηρίζουμε την προσχωρική στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις διάφορες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και με την σύνδρομη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλους δωρητές. Εμείς θέλουμε να διπλασιάσουμε τα κονδύλια που δίδουμε για την περιοχή, πράγμα που σημαίνει ότι φέτο αυτός από 18,5 ε, θα δοθούν περίπου 37 εκατομμύρια ευρώ του χρόνου. Για επίσης θέλουμε να μπορέσει να προωθεί η οικονομική συνεργασία, η καλή διακυβέρνηση, η καταπολέμηση της διαφθοράς του οργανωμένου κλίματος και τα βελτίωση των κοινωνικών συνθήκων. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει τα διάφορα κονδύλια να δημιουργήσουν συνθήκες ε, θετικές σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι υποφελές όχι μόνο για τις χώρες της περιοχής αυτής, αλλά ε, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι μακροπρόθεσμα ο στόχος είναι να γίνει οικονομικά όλο και λιγότερο εξαρτημένη η περιοχή. Πιστεύω ότι εμείς ε, με τα βοήθειά μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε την περιοχή αυτή και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθούν κονδύλια όπως σας είπα και από εμά τα επόμενα ε, νέα χρόνια στα πλαίσια ενός νέου Ταμείου Συνεργασίας 35 νέα ε, εκατομμύρια ώστε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε σχέδια ανάπτυξης περιοχής. Θα ήθελα να πω ότι για να είναι επιτυχές οποιοδήποτε ε, πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει μόνο όταν δεν υπάρχουν περαιτέρω ε, διανέξεις και φιλονικίες ε, και μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων. Ευχαριστώ. Παίρνουμε τώρα στην κυρία Ροζαλία Μπύρου από τη Ρουμανία. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή και ευκαιρία για εμάς που βρισκόμαστε εδώ Γι' αυτόν τον διάλογο. Θα συνεχίσω τώρα στην Ρουμανική. Εμείς υποστηρίζουμε την πολιτική διεύρυνση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τις προσπάθειες που κάνουν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θεωρούμε ότι είναι μια γεωπολιτική προτεραιότητα και είναι κλειδί για την σταθερότητα, την ειρήνη και την ευμερία στην περιοχή. Οι προοπτικές ε, για την Άνοιξη 2018 είναι πάρα πολύ καλές. Η Βουλγαρική Προεδρία θα οργανώσει μια σύνοδο κορυφής σε ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον, αλλά η κατάσταση είναι περιπλοκή και θα πρέπει να βοηθούν οι χώρες ε, στην πορεία των μεταρρυθμίσεων. Η Ρουμανία θα ήθελε να υπάρχει ένας μόνιμος διάλογος με αυτές τις χώρες και να τις βοηθούμε Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας για να ενισχύσουμε και τις δημιουργίες μας σχέσεις με τις χώρες αυτές. Μπορούμε νομίζω να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων και να δώσουμε πιο ουσιαστικές απαντήσεις στις προσδοκίες τους και στις χώρες μας και στις χώρες αυτές. θα προετοιμαστούμε εμείς για την ε, δική μας ε, Προεδρία του Συμβουλίου και θα θέλαμε ακριβώς να έχουμε μια διαβριμένη ένωση με κοινές αρχές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα δίνω τον λόγο στον Γιώζεπ Γιμποράτοβιτς από την Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που διαπιστώνουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε τα Δυτικά Βαλκάνια όπως και αυτά μας χρειάζονται για λόγους ασφαλείας. Η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια δεν είναι υποδειγματική. Θα έλεγα υπάρχουν... Υπάρχει ένα πολιτικό κλίμα, οι χώρες οι οποίες κέρδισαν τον πόλεμο δεν βιάζονται και να ενταχθούν. Αλλά υπάρχουν και θετικές εξελίξεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί που ζουν το ευρωπαϊκό πνεύμα. πολιτικοί, νέοι, διανοούμενοι, οι οποίοι κάνουν επαφές διασυνοριακές, ε, συμμαχίες, ε, επιχειρηματίες και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι μπορούν δυστυχώς να χαρακτηριστούν ως νοσταλγοί της ε, Ιουγκοσλαβίας. Θα πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους ε, που έχουν ευρωπαϊκό πνευμά. Δυστυχώ ε, είναι γεγονός πως στα Δυτικά Βαλκάνια θα έλεγα ότι συνολικά έχουμε μια ανεργία των νέων γύρω στο 50%. Πάρα πολλοί νέοι καταφεύγουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχει και η άλλη πτυχή που διαφθείρει ή ριζοσπαστικοποιεί τους νέους. Γι' αυτό χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη, γι' αυτό χαιρετίζω την διαδικασία αυτή του Βερολίνου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο για την ένταξη και την σταθεροποίηση της περιοχής. Επίσης, η, διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει και μια διαδικασία ένταξης, γιατί βεβαίως, πρέπει η ανάπτυξη να συνοδευτεί από καταπολέμηση της διαφθοράς και εκδημοκρατισμή. Δηλαδή, εάν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την διαφθορά, θα πρέπει να στηρίξουμε και οικονομικά αυτήν την περιοχή. Βεβαίως δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος αυτοματισμός όσον αφορά τα 35 κεφάλαια. Πρέπει να εφαρμοστούν, όχι μόνο να νομοθετηθούν, αλλά να γίνουν πράξη. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μένα να αναφέρω είναι ότι ε, είναι δύο χώρες, ε, δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλες, ε, κυρίως να αναφερθώ στη Μακεδονία και την Βοσνία Ζεγοβίνη. Για εμάς η Μακεδονία είναι η λιδία λίθος της αξιοπιστίας. Θα το πω ξεκάθαρα. Το κίνημα αυτών των πολιτών του εκδημοκρατισμού πρέπει να στηριχθεί επιγόντως ε, και βεβαίω η δικαιολογία περί ονόματος που χρησιμοποιούμε ε, πρέπει να παραμεριστεί. Πρέπει λοιπόν και να εργαστεί από αυτού του προβλήματος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον για την Βοσνία Ζεγοβίνη, ε, δύο χώρες είναι πολύ σημαντικές, η Σερβία και η Κροατία, που έχουν υπογράψει την συμφωνία του Dayton και έχουν υποχρεώσεις ε, να μην στηρίζουν δηλαδή την δική τους εθνότητα αλλά την χώρα στο σύνολό της για να υπάρξει εκδημοκρατισμός. Και τέλος είναι πάρα πολύ σημαντικό στη Σόφια και στη Βουλγαρία να έχουμε μία πολιτική ε, η οποία θα δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα έργο ειρήνης και όχι μόνο μία αγορά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γιουράτοβιτς και σας ευχαριστώ που εκπροσωπείτε την περιοχή αυτή στην Γερμανική Βουλή. Περνάμε τώρα στον επόμενο μιλητή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Νίνο Μπιτσουλά από την Κροατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να παραθέσω τον κύριο Ντάνιουσον που παρέθεσε τον κύριο Γιούνκερ. Σαφή προοπτική για την Ευρώπη, για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Το πλαίσιο κρίση των διαπραγματεύσεων ελέγχθη ότι θα είναι το 2025. Πριν από μερικά χρόνια στην Σύνοδο Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε η προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλων των ε, ε, χωρών των Δυτικών Βαλκίων. Μέχρι τώρα μόνο εμείς στην Κροατία το καταφέραμε. Βεβαίω, όλα εξαρτώνται το πώ βλέπει το μέλλον τη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είδου Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε μετά την επόμενη διεύρυνση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα όπως η οικονομική κρίση από το 2008 και μετά και διερωτάται πώς θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα θέματα της ασφαλείας είναι το πρωταρχικότερο θέμα που μας απασχολεί. Αλλά πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο σε τέτοιου είδου προβληματισμό μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκονται κοντά στην περιοχή στην οποία υπάρχει σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Το 2015 κάποια στιγμή η μεταναστευτική κρίση πρέπει να πω ότι ξανάφερε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο προσκήνιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη. Και βεβαίως εκεί τέθηκε θέμα σταθερότητας και ασφάλειας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι άμεση γείτονε, αλλά είναι στα εσωτερική αυλή μας οι χώρες αυτές. Επίσης, σύντομα, θα πρέπει να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα. Η δημοκρατία δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την σταθερότητα στην περιοχή. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε Προσεκτική, ώστε να έχουμε τους ε, κατάλληλους ηγέτες που θα δώσουν τεν, στους πολίτες δυνατότητες ανάπτυξης και θα είναι υπέρ του πολιτικού ε, πλουραλισμού. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ζαμπιέρο Ζουάνα. From Italian Parliament από την Ιταλική Βουλή. Sí. Τον κύριο Ζαμπιέ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας από την Ιταλική Γερουσία. Παίρνω το λόγο ως πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής για την ε, ομάδα φίλων ουσιαστικά με το κοσφοπέδιο. Δύο-τρία πράγματα θέλω να πω μόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το κοσφοπέδιο να αναγνωρίσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το έχουν πράξει ακόμα το κράτος αυτό. Και θα πρέπει βέβαια και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει διπλωματική πίεση προς τις χώρες εκείνες του κόσμου τώρα που δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα το κοσφοπέδιο. Αυτό παράλληλα με μια πλήρη οικονομική ολοκλήρωση της χώρας αυτής και μια υποστήριξη προς το κοσφοπέδιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δεν είναι θετικό ότι το Σεπτέμβριο για μία ακόμα φορά απορρίφθηκε το αίτημα προσχώρησης του Κοσφοπεδίου στην Ίντερπόλα. Μιλάμε για παγκόσμια συνεργασία για την καταπολέμηση τρομοκρατίας και δεν μπορούμε καν να παραχωρήσουμε προσχώρηση του Κοσφοπεδίου στην Ιντερπόλ. Κάτι ακόμα τώρα, όσον αφορά τις θεωρήσεις. Σίγουρα το πρόβλημα του κοσφοπεδίου και των θεωρήσεων δεν αφορά μόνο το κοσφοπέδιο, αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ε, δεκάδες ε, χιλιάδες, 40.000 ε, περίπου για παράδειγμα κάτοικοι του κοσφοπεδίου μόνο και μόνο στην Ιταλία και ουσιαστικά ένα 2-3% της χώρας βρίσκεται ήδη στην Ιταλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να προχωρήσουμε στην απελευθέρωση των θεωρήσεων για να απαλλάξουμε τους ανθρώπους αυτούς από το τεράστιο αυτό γραφειοκρατικό άχθος, αλλά όχι μόνο τους πολίτες του Κοσυφοπεδίου, αλλά και τις ίδιες τις διοικητικές αρχές της χώρας αυτής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντας λοιπόν γερουσιαστής που συμμετέχει στην ομάδα φιλίας με το Κοσμοπέδιο, θεωρώ ότι τα σημεία αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν σημεία επί των οποίων θα σημειώσουμε πολύ σύντομα πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόοδο αυτή θα είναι θετική τόσο για εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για το ίδιο το Κωσυφοπαίδιο. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Ζωάνα. Το λόγο τώρα έχει ο κύριο Δημήτρος Εμμανουλίδη από την Ελλάδα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η προοπτική περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως η προοπτική ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ένωση αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ελλάδας. Φυσικά από πλευρά των κρατών αυτών πρέπει να εκπληρώσουν όλα τα κριτήρια της Κοπενχάγης και των υπόλοιπων προαπαιτούμενων. Το κοινό μας μέλλον στα Βαλκάνια δεν μπορεί να κτιστεί πάνω στον εθνικισμό όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Δεν μπορεί να χτιστεί ούτε σε σχεδιασμούς τρίτων για την περιοχή μας. Μπορεί να χτιστεί μόνο στις μεγάλες δυνατότητες των λαών μας, στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σε ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα για την περιοχή μας. Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Βαλκανίων πρέπει να είναι μια πορεία που βασίζεται σε ένα νέο όραμα για τη συνεργασία λαών στην ευρύτερη περιοχή. Τα Βαλκάνια είναι μια πολύ κρίσιμη περιοχή για την Ευρώπη. Είναι μια περιοχή που στο παρελθόν γέννησε πολέμους και αντιθέσεις. Σήμερα όμως μπορεί να γεννήσει την ελπίδα για μια νέα πορεία συνεργασίας και συνανάπτυξης. Η ευρωπαϊκή προοπτική συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή. Υποστηρίζουμε την ενταξιακή πορεία της ΦΥΡΟΜ έχοντας συμβάλει ενεργά στην προώθησή της σε πολλά κρίσιμα σημεία. Τονίζουμε όμως παράλληλα τη σημασία εκπλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων και προαπαιτουμένων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο ζήτημα του ονόματος, καθώς και την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπενχάγης. Υποστηρίζουμε επίσης την ενταξιακή πορεία της γείτονος Αλβανίας, σημειώνοντας την ανάγκη περαιτέρω προσπαθειών σε κέρυες προτεραιότητες. Αυτές αφορούν τόσο τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήματος, όσο και την ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση των διακρίσεων περιλαμβανομένων των μειονοτήτων όπως αναφέρουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 15 12 του 2015, υπάρχει ανάγκη της ίσης μεταχείρισης όλων των μειονοτήτων και πρόσβαση στα δικαιώματά τους σε όλη την επικράτεια της Αλβανίας καθώς και την, της εφαρμογής των περιουσιακών δικαιωμάτων. Η χώρα μας παραμένοντας σταθερή στην ανάγκη διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων υποστηρίζει την ενταξιακή τους πορεία με την προϋπόθεση βέβαια να τηρηθούν από τις ενδιαφερόμενες χώρες οι δεσμεύσεις που υπαγορεύονται από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στο κράτος δικαίου και στις σχέσεις καλής γειτονίας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. A sada ću Branku iz Crne Gore da nam se σας ευχαριστώ κυρία Μπάνκα Ντάν από το Μαυροβόνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη τιμή συμμετείχα στη συνεδρίαση αυτή και εκπροσωπώ το Μαυροβούνιο που έχει επιτελέσει μεγάλη πρόοδο. Πράγμα το οποίο ελέγχθηκε χθε στην συνεδρίαση των Αγγελής Τραπέζης. Θα ήθελα επίσης να πω ότι οι δυνατότητες και οι δεσμεύσεις των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων διαδραματίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την ένταξή τους στην Ευρώπη. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και τη θέση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποστήριξη των κρατών μελών για την προσχώρηση των, Δυτικών Βαλκαν... χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. εδώ και λίγο καιρό έχουμε όλο και πιο σαφή μηνύματα όσον αφορά την προσχώρηση. Και το μήνυμα της ε, συνεδρίασης θέση ήταν εξίσου σαφής με αυτό του Πρόεδρου Γιούγκερ όσον αφορά την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μήνυμα το οποίο επιβεβαιώνει τις προσπάθειες που γίνονται υπέρ της συνοχής. Όταν ε, επίσης ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Μακρόν στη Σορβόνη είπε ότι θα πρέπει να μπουν σε πρώτη προτεραιότητα οι προσπάθειες περαιτέρω διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική λοιπόν της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής που θα δημοσιευτεί τον Φεβρουάριο θα δώσει μια νέα πρόπτικη στην προσχώρηση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Το 2025 δεν θυμαίνει ότι η προσχώρηση θα πρέπει να γίνει απαραίτητο το 2025. Αν κάποια χώρα είναι έτοιμη πριν, θα πρέπει να είναι έτοιμη να την υποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως αναφέρομαι στο Μαυροβούνιο, το οποίο έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό πάρα πολλές προσπάθειες στον ε, οικονομικό τομέα και σε άλλους. Επίσης, με την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ, η στρατηγική δικές μας επιλογές ε, επιβεβαιώθηκαν και μετά από την ε, ανεξαρτησία μας πριν από περισσότερο από 10 χρόνια έχουν επιβεβαιωθεί αυτά που λέω. Αυτό που λέω για τη χώρα μου ε, ίσως ισχύει και για άλλες χώρες και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το Μαυροβούνιο θα υλοποιήσει όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στα πλαίσια της προσχώρησης. Έχουμε ανοίξει 28 κεφάλαια, έχουμε προσωρινά κλείσει τρία και για τα υπόλοιπα είμαστε διατεθειμένοι να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες περιμένοντας και να ανοίξουν και νέα κεφάλαια τους επόμενους μήνες. Επίσης, είμαστε υπέρ της λήψης συμπληρωματικών μέτρων, κυρίως σε θέματα κράτους δικαίου, παρά το γεγονός ότι ήδη έχουμε κάνει πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Συμπερασματικά θα πω ότι η πρόεδρος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εμά, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι και τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα είναι αυτά τα οποία καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα σε σχέση με τα συμφέροντά τους και τις στρατηγικές τους. Κατά συνέπεια, ένας νέος δυνασμισμός στις περαιτέρω εξελίξεις θα μας οδηγήσει στο να ολοκληρώσουμε έγκαιρα τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρκ Ογκλού από το Λουξεμβούργο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσω και με τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά από και τα κοινοβούλια των Δυτικών Βαλκανίων. Η δεύτερη συνεδρίαση που συμμετέχω είναι αυτή. Ο Επίτροπος Μίμητσα σήμερα το πρωί αλλά και σήμερα το απόγευμα ο Επίτροπος Χάν υποτίθεται ότι θα μιλούσαν. Είναι κρίμα που δεν ήρθαν τελικά γιατί θα ήταν πολύ σημαντικό τους είχαμε εδώ πέρα και να συζητούσαμε και μαζί τους. Παρόλα αυτά Πρέπει να πω ότι εκτίμησε ιδιαίτερα τα όσα μας είπε ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Κρίστιαν Ντάνελσον, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο ζήτημα της συμφιλίωσης, που θεωρώ ότι πραγματικά μπορεί να αποτελέσει πυλώνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφιλίωση, να θέλετε, το καλύτερο φάρμακο κατά του εθνικισμού. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους από τα Δυτικά Βαλκάνια, από τα κοινοβούλια των Δυτικών Βαλκανίων, ότι το Λουξεμβούργο, η χώρα μου, υποστηρίζει τη διαδικασία προσχώρησης των χωρών του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορά στη συζήτηση που γίνεται στα πλαίσια των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δικός μου Υπουργός, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και όταν έρχεται στη δική μου την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, της οποίας προεδρεύω, μιλάει πάντα θετικά υπέρ της διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Εκτιμώ επίσης πάρα πολύ το νέο μήνυμα που προωθεί πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νέο σλόγγαν Fundamentals First, πρώτα τα θεμελιώδη ζητήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, όντω να επικεντρωθούμε στα κεφάλαια 23 και 24. Τα θεμελιώδη αυτά σημεία βέβαια είναι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και ξέρουμε επίση και ότι οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών είναι οι καλύτεροι υποστηρικτές και οι καλύτεροι, αν θέλετε, παράγοντες μπορούν να παρακολουθήσουν την ε, έμπρακτη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Ζητάνε ελευθερία του τύπου, ελευθερία της έκφρασης, περισσότερη διαφάνεια και δεν φοβούνται να θίξουν ζητήματα όπως η διαφθορά. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι στα πλαίσια του μηχανισμού προταξιακής βοήθειας. Θεωρείτε ότι κάνουμε αρκετά πράγματα εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτώντας ε, την κοινωνία των πολιτών στα Δυτικά Βαλκάνια η χρηματοδότησή μας και η γενικότερη υποστήριξή μας προς τα Δυτικά Βαλκάνια ομοιάζει με την υποστήριξη που δίνουμε προς την κοινωνία των πολιτών στην ανατολική εταιρική σχέση. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Πώς αξιολογείτε εσείς την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες σας στα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε τώρα στον επόμενο ομιλητή, την κυρία Ρουμάνα Γέρκοβιτς από την Κροατία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας μιλήσω και να ανταλλάξω με σας απόψεις για το σημαντικότατο αυτό ζήτημα, προσχώρηση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με τα όσα είπαν οι κύριοι Κόβατς και Πίτσουλα από την Κροατία. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται για να πω για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η προσχώρηση αυτή των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων για τη χώρα μου την Κροατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνειδητοποιήσει, θεωρώ, πόσο πολύπλοκη είναι η διαδικασία της διεύρυνσης. Πρόκειται για μία μακρόπονη διαδικασία, που επηρεάζεται όμως και από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καταλήγουμε τελικά σε έναν κίνδυνο. Ένα κίνδυνο τον οποίο τον αναφέραμε και στην αρχή της συνεδρίασης αυτής. Ο κίνδυνος είναι να οπισθοδρομήσουμε τελικά και να χάσουμε τον δυναμισμό αυτόν τον οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τώρα να προωθεί περισσότερο και να υποστηρίζει περισσότερο την ενταξιακή προοπτική των χωρών αυτών. Και θα πρέπει μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ρόλο πρωτοπόρου, να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της υποστήριξης των χωρών αυτών, να καταφέρει να επηρεάσει θετικά τα Δυτικά Βαλκάνια και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να επικεντρώνεται στο ζήτημα της διεύρυνσης αφού είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη βέβαια. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλεγε χώρα το Μάρτιο. Να χαιρετήσω επίσης ε, το λόγο του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, κ. Γιούγκερ που είπε ιδιαίτερα θεραντικά λόγια όσον αφορά την προοπτική διεύρυνση των χωρών αυτών. Βλέπουμε πλέον ότι τα λόγια αρχίζουν και αντιστοιχούν περισσότερο σε πράξεις και θα ήθελα να έλεγα στον, επίτροπο, στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούνκερ ότι έχω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στα όσα λέει και θα ήθελα βέβαια να ελοποιηθούν πλήρω στην πράξη. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις πολύ αυστηρές αλλά δίκαιες προϋποθέσεις που έχουμε θέσει όσον αφορά την ενταξιακή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν μπορούμε βέβαια να περιμένουμε μία νυχτή να γίνουν θαύματα. Η πρόοδος πιστεύω ότι θα λάβει χώρα αργά ή γρήγορα χάρη στην προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταβάλουν ακόμα περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να στηρίξουν τις χώρες του Δυτικών Βαλκανίων και να τους δώσουν τα απαραίτητα κίνητρα για να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου, τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού, δικαστικού συστήματος. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Έχουμε τώρα νομιλητή από την Πορτογαλία, Βιταλίνο Κάρνιας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχίζοντας να υπογραμμίσω ότι με εντυπωσιάζει ο ενθουσιασμός των εκπροσώπων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που ήρθαν εδώ να παρουσιάσουν την ε, ευρωπαϊκή τους προοπτική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την εσωτερική μας πολιτική συζήτηση. Μόνο που είμαστε ήδη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρουμε ότι στις χώρες μας κάποιοι πολίτες αρχίζουν να έχουν μία στάση σκεπτισμού όσον αφορά την ε, Ευρώπη. Και όταν ακούμε το, με τόσο ε, ενθουσιασμό και τέτοια δυναμική της παρεμβάσης των συναδέλφων, πιστεύουμε ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι το σημαντικό και γι' αυτό το τονίζω. Μου φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα θα πρέπει να δώσουν την δέουσα σημασία σε αυτό το γεγονός. Πολλές φορές οι πολιτική δεν είναι απλώς η εκτίμηση των συγκυριακών συμφερόντων. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πολλές φορές και ο ενθουσιασμός και το πάθος κάποιου για μια κατάσταση. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει λοιπόν να μην είναι θετική προς αυτή την προσέγγιση των ε, χωρών Δυτικών Βαλκανίων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες εκ μέρους κάποιων κρατών, εκ μέρους των κρατών που θέλουν να προσχολήσουν, αλλά θα ήθελα να κάνω δύο γενικής ω σχόλια. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να κάνω έκκληση ώστε οι χώρες αυτές να αντισταθούν σε κάποιους πειρασμούς που αντιμετωπίζουν και με την δική μας συνδρομή και να καταλάβουν ότι κάποιοι παίκτες εκτός Ευρώπης προσπαθούν όπως είπα και εκείνα να παίξουν σημαντικό ρόλο στη χώρα τους και τους λένε ένα πάρα πολύ μελωδικό τραγούδι αλλά θα πρέπει να αντισταθούν. Η προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει χωρίς καθυστερήσεις. Δεν θα γίνουν οι καθυστερήσεις, δεν θα μπορέσουν να προσχωρήσουν έγκαιρα. Επίσης, πιστεύω ότι οι μεταρρυθμίσεις που ζητούν δεν θα πρέπει να γίνουν εκ μέρους των χωρών αυτών κατανοητές ως κάτι το επιτακτικό. Πρόκειται για σημαντικές και θετικές μεταρρυθμίσεις για τις χώρες αυτές, για τους πολίτες των χωρών σε όλους τους τομείς, τη δικαιοσύνη μεταξύ άλλων. Και δεν ε, είναι θέμα ε, προσέγγισης όλο και περισσότερο της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να οδηγήσει τις χώρες αυτές στο να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος Γιούγκερ. Συμφωνώ απόλυτο και νομίζω ότι κάθε χώρα που θα ε, μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραμμά της και να ε, ικανοποιήσει τα κριτήρια και τα προαπαιτούμενα, θα πρέπει να προσχωρεί και να μην περιμένει και τους άλλους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στον κύριο Φρουντζουλίκα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Μάλιστα, πρόσφατα είδα κάποιες δηλώσεις ηγετών της Ένωσης που θεωρούσαν τα Δυτικά Βαλκάνια ως μια προβληματική γείτονια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι λάθος. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι στο κέντρο της Ευρώπης και πρέπει να επιταχύνουμε την ένταξή τους. Είναι μια σημαντική και στρατηγική περιοχή της Ευρώπης και δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε μια τέτοια ζώνη ως ένα κενό, ως μια γκρίζα ζώνη στην Ευρώπη. Και πρέπει μετά το Brexit να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ε, διεύρυνση και να έρθουμε ξανά σε επαφή με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, γιατί η κατάσταση χειροτερεύει. 43% των πολιτών των Βαλκανίων έχουν σκοπό να μεταναστεύσουν αλλού, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη. Η ανεργία των νέων είναι υψηλότερη στην Ευρώπη. Παραδείγματο χάρη στην Βοσνία Ζεγοβίνη 56%, 39% στο Μαυροβούνιο. Δυστυχώ η στήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται. 39% του κοινού δεν θεωρούν πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι καλό για την οικονομία τους. Χρειάζεται λοιπόν, πρέπει να πούμε στα ευρωπαϊκά θεσπικά να, να ξεκινήσουν μια νέα στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια, γιατί η κατάσταση χειροτερεύει. Βλέπετε νέες εθνοτικές εντάσεις με την κατάσταση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρη για αυτές τις χώρες. Έχουμε νέες δηλώσεις από το Κοσφοπόδιο για το Μαυροβούνιο, η... από την Σερβία για το όνομα της Μακεδονίας ή από την Αλβανία που μιλάει για αλβανικές ε, περιοχές ε, γύρω από την Αλβανία. Και οπωσδήποτε ε, και πρόεδρε, πρέπει να οδηγηθούμε σε μια διαδικασία Βερολίνου συν να εφαρμόσουμε μια νέα στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκανία γιατί έχουμε ε, μια στασιμότητα, ναι, μια διαδικασία Βερολίνου, να βελτιώσουμε τη διασύνδεση, δηλαδή μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι παραπάνω, γιατί αν συνεχίζουμε ε, επί χρόνια, έτσι, ο κόσμος των Δυτικών Βαλκανίων δεν θα ε, θεωρεί πια ότι το μέλλον τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είναι η στιγμή να αλλάξουμε υπόδειγμα στα Δυτικά Βαλκάνια, να βρεθεί μια νέα στρατηγική γιατί το μέλλον τους είναι στην Ευρώπη, όχι σε άλλες χώρες που θέλουν να αυξήσουν την ε, επιρροή τους και την οικονομική τους ε, εμπλοκή εκεί. Η χώρα μου, η Ρωμανία, στηρίζει, όπως ξέρετε, την ένταξη όλων αυτών των χωρών και των έξι χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ξεκινήσουμε ε, γρηγορότερα από ότι νομίζαμε πριν από λίγα χρόνια ότι που λέγαμε ότι δεν θα έχουμε νέο κράτος μέλος τα επόμενα πέντε χρόνια. Πρέπει να ξεκινήσουμε με μία-δύο χώρες και να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Φρουντσουλίκα. Ε, κατάλαβα καλά τώρα έχουμε τον τελευταίο μιλητή που έχω στον καταλογό μου, ο κύριος Ζόλτ Ζάλαν. Κάποιος άλλος θέλει τον λόγο, όχι, κλείνει. Λοιπόν, ο κατάλογος των μιλητών, Ζόλτ Ζέγκερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά την Ουγγαρία, μας ενδιαφέρει και είμαστε προσιλωμένοι στην διεύρυνση. Είναι ηθικό μας καθήκον, θα έλεγα, και είναι ηθικό καθήκον, γιατί επί σειρά ετών οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ε, κατέβαλαν εξαιρετικές ε, προσπάθειες για να ενταχθούν και βέβαια μιλάμε για τους ανθρώπους ε, επιτόπου που έκαναν τεράστιες θυσίες. Αλλά δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση, είναι νομίζω και ένα ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για εμάς. Η σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας ε, όσον αφορά την σταθερότητα και την ασφάλεια. Είναι σημαντικό για την Ευρώπη, για την ευρωατλαντική περιοχή. Πρέπει να εντάξουμε αυτές τις περιοχές το στομότερο δυνατόν. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην περιοχή επειδή έχει καθυστερήσει η διαδικασία διεύρυνση και βεβαίω αυτό επηρεάζει τρίτες χώρες. Υπάρχουν άλλες χώρες που θέλουν να γεμίσουν αυτό το κενό. Οπότε θα πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις χώρες γιατί εάν δεν το κάνουμε θα το κάνουν άλλοι. Και αυτό πρέπει να το αποτρέψουμε. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ το ανέφερε αυτό. Είπε ότι η διεύρυνση είναι σημαντική και πρέπει να στηριχθεί. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει την διαδικασία διεύρυνσης και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με την Κομισιόν στην επεξεργασία των στρατηγικών εγγράφων. Χρειαζόμαστε επίσης ένα χρονοδιάγραμμα σε σχέση με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο και να πούμε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος και να ακολουθούμε και εμείς όσο προχωρούν αυτές ε, όσον αφορά την Αλβανία. Πρέπει να δοθεί η ημερομηνία. Βοσνία Ζεγοβίνη, Κοσμοπέδιο. Ελπίζω να έχουν κάποιους εφικτούς στόχους στο προσεχές μέλλον και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ΝΑΤΟ. Μπορεί το Δεκέμβριο να προκύψει το θέμα της Μακεδονίας και κάποιες επίσημες διαπραγματεύσεις. Επίσης, Βοσνία Ζεγοβίνη υπάρχει το σχέδιο ένταξης ε, όσον αφορά λοιπόν την Ουγγαρία, η εξωτερική μας πολιτική ήταν επιτυχής. Ε, πρόσφατα, παραδείγματο χάρη, να αποφασίσαμε να αποστείλουμε συμβούλους ε, στο Βελιγράδι, στα Τύρανα, στην Ποντγκόριτσα και αλλού. Στέλνουμε λοιπόν αυτούς τους εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να προετοιμαστούν για την ένταξη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ χρήσιμο και θα κάνουμε κάτι ανάλογο για το κοσυφοπέδιο. Όπως σας είπα λοιπόν είναι προς το συμφέρον της Ουγγαρίας ε, να ενταχθούν αυτές οι χώρες το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τα σχόλιά σας. Ναι, κάλυψαν ένα ολόκληρο φάσμα από ερωτήσεις μέχρι δηλώσεις. Νομίζω πως οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούσαν τον κύριο Ντάνιλσον. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτόν και μετά να δώσουμε τον λόγο στην ε, κυρία Άιχοστ και τέλος ε, στην κυρία Πέντους Ροζημάνους και τον κύριο Κρίστο από την Βουλγαρία και ο Ντουαρτ Κούκαν ε, έχει φύγει. Λοιπόν, Ξεκινάμε με τον κύριο Ντάνιελσον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις, τις δηλώσεις και τις ερωτήσεις σας, ιδιαίτερα επικοδομητικές και χρήσιμες, διότι βρισκόμαστε στην διαδικασία της επεξεργασίας της μελλοντική αυτής στρατηγικής που θα παρουσιάσουμε το Φεβρουάριο του 2018. Πολλές λοιπόν ιδέες και σκέψεις ακούστηκαν, οι οποίες πραγματικά εμπλουτίζουν την όλη διαδικασία. Είναι σαφές από ευρωπαϊκής πλευράς, από τα όσα ακούσαμε σήμερα εδώ πέρα, ότι επιβεβαιώνεται εκ νέου η σημασία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και είναι σημαντικό να επανεπιβεβαιώσουμε την προοπτική της ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, προκειμένου η προσχώρηση των κρατών αυτών να αποτελέσει πραγματικότητα και νομίζω ότι πολλοί το είπαν αυτό και όχι μόνο οι βουλευτές από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Και πολλές από τις μεταρρυθμίσεις αυτές ήδη έχουν ξεκινήσει, πολλές έχουν ήδη εφαρμοστεί. Αυτό που φάνηκε όμως από τη συζήτηση περαιτέρω είναι ότι δεν αρκεί να αναφερόμαστε γενικά και αόριστες μεταρρυθμίσεις ή απλώς αυτές να εγκρίνονται από τα κοινοβούλια, αλλά θα πρέπει και στην πράξη να εφαρμόζονται. Και βέβαια συνδέονται με τα κριτήρια της Κοπενχάγης, τα οποία αναφέρθηκαν, αλλά σχετίζεται το ζήτημα αυτό και με την μελλοντική μορφή που θα έχουν οι κοινωνίες από τις χώρες αυτές και αναφέρεται επίση και στη δυνατότητά τους να οδηγηθούν στην απαραίτητη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν και από τους προαλήσαντες ιδίω για να πατάξουμε αρνητικά φαινόμενα όπως η ανεργία των νέων ή προκειμένου να έχουμε ευίωνες οικονομικές προοπτικές για το μέλλον. Και θα πρέπει βέβαια όλη αυτή η διαδικασία να είναι πλαισιωμένη και εδώ έρχονται να δραματίσουν σημαντικότατο ρόλο τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μελών, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που θα πρέπει από κοινού να συνεργαστούν για την παροχή συμβουλών αναπόσπαστο τμήμα αυτό της όλης διαδικασία να είναι σε θέση επίση να δείχνουν κάθε φορά τι πρέπει να γίνει για να ανταποκριθούν οι χώρε αυτέ αυτές τις προσδοκίες μας, αλλά να παρέχουν και τα απαραίτητα συνοδευτικά μέτρα προκειμένου να μπορούν όντω οι χώρε αυτέ να ταπεξέλθουν στι απαιτήσει μα. Και αναφέρομαι στην χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη και στα συναφή και τέθη ω προς αυτό και ένα ερώτημα όσον αφορά την υποστήριξη προς την κοινωνία των πολιτών. Λοιπόν, ως προς αυτό σας επιβεβαιώνω ότι όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, προσπάθειες τι οποίες προφανώς στηρίζουμε, το ζήτημα της κοινωνίας των πολιτών είναι κομβική σημασία. Γι' αυτό το λόγο η στήριξη που δίνουμε προς την κοινωνία των πολιτών είναι και θα συνεχίσει να είναι θεμελιώδου σημασίας. Μια τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Είναι ένα ερώτημα ουσιαστικά που ετέθη. Ο εκπρόσωπος της, ή εκπρόσωπος μάλλον της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης αναφέρθηκε στο ζήτημα των συστάσεων προς την Αλβανία και την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αν κατάλαβα καλά πότε θα γίνουν αυτές οι συστάσεις, πότε να τις περιμένουμε, μας ζητήσατε. Σα διαβεβαιώ ότι από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπής εμείς θα προχωρήσουμε στις συστάσεις αυτές μόλις δούμε ότι τα κριτήρια τα οποία έχουμε θεσπίσει όλα αυτά τα οποία θέλουμε δηλαδή να δούμε να γίνονται και να ελοποιούνται στις χώρες αυτές και στις εκθέσεις προόδου από το Δεκέμβριο του 2015 και μετά έχουμε αποσαφηνίσει όλα αυτά τα κριτήρια προς όλες αυτές τις χώρες. Αυτή τη στιγμή αρχίσουν να πληρούνται τα κριτήρια αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας βεβαιώ θα προχωρήσει σε επίσημες συστάσεις. Δεν έχουμε φτάσει όμως ακόμα στο σημείο αυτό. Μας ενθουσιάζει πραγματικά η όλη ιδέα ότι οι χώρες αυτές πλησιάζουν στη φάση αυτή, η οποία όμως δεν έχει έρθει ακόμα. Τούτων λεχθέντων ολοκληρώνω στο σημείο αυτό και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσετε να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση, η οποία ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική. Σα ευχαριστούμε κύριε Ντάνιελσον και εμεί σα ευχαριστούμε γιατί η παρουσία σας εδώ πέρα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και βασιζόμαστε και στην περαιτέρω υποστήριξή σας στο μέλλον. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Άιχόρστα. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, να απαντήσετε σε κάποιε ερωτήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη που συμμετείχαν στην εξαιρετική αυτή συζήτηση. Δύο παρατηρήσεις. Ξέρουμε ότι πρέπει να επιτελεστεί μεγάλη δουλειά. Το γνωρίζουμε όλοι. Νομίζω ότι πρόκειται για μία διαδικασία η οποία θα πρέπει να γίνει με συνεκτικό, επικοδομητικό τρόπο και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι. Συνεκτικότητα, συνοχή και με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να εργαστούμε και να προχωρήσουμε με ρεαλιστικό τρόπο και να δώσουμε τα σωστά μηνύματα σε όλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μέρος της στρατηγής μας να δίδουμε, να δίδονται μηνύματα σε όλο τον κόσμο στην περιοχή αυτή με σαφήνεια. Όλα αυτά γίνονται με προσόφελες και των πολιτών των χρόνων αυτών και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόλυτη σαφήνεια λοιπόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Από τη δική μας την πλευρά συμπεριλάβαμε τις υποψήφιες χώρες σε διάφορες διαδικασίες που αναλαμβάνουμε στα πρέσια της Προεδρίας. Το Δεκέμβριο οι Υπουργοί των Υποψηφίων Χωρών έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση που θα έχουμε με την παρουσία του Επιτρόπου ΧΑΝ στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Αυτού του είδους η συνεργασία θετικά είναι εξαιρετική και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόμη μια φορά να επαναλάβω ότι σήμερα έχουν αναφερθεί πολλές ευκαιρίες που θα χρησιμοποιηθούν από του χρόνου. Εμείς είμαστε από τη μεριά μας πεπισμένοι ότι η επόμενη Προεδρία της Βουλγαρίας που θα ακολουθήσει τη δική μας θα εστιαστεί και εκείνη στα θέματα της προσχώρησης των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Και τώρα φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι τις προσπάθειες που κάνετε ώστε με διαφάνεια να προοδεύσετε ώστε να υπάρχει προσχώρηση των κρατών αυτών. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το απεφελές και για σας και τις χώρες της και για μας. Όπως ξέρετε οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν διανύσει μεγάλη απόσταση μέχρι σήμερα. Τώρα θα πρέπει να γίνουν τα τελευταία βήματα για να φτάσετε στο τελικό σημείο της προσχώρησης, για την προσχώρησή σας. Ξέρω ότι κάθε περίοδος είναι περίοδος προκλήσεων σε σχέση με την προηγούμενη, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να, να προωθήσουμε την ελευθερία, τη δημοκρατία, τη σταθερότητα και οι κοινωνίες μας νομίζω ότι εκτός από την κοινωνική ανάπτυξη θα πρέπει να βλέψουν και στην ευημερία. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις για όλους, αλλά θα πρέπει μέσω κοινών ε, προσπαθειών να βελτιωθεί η διακυβέρνηση, η συνεργασία στην περιοχή και να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υποστηρίζει την ε, μακροχρόνια ευημερία των λαών των χωρών σας. Να μην ξεχνάτε ότι η προσχώρησή σας είναι ένα βήμα ακόμη προς την θεμελίωση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεισφορά σας στην ανταλλαγή απόψεων και προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία μεταξύ ημών και ημών.